Ας αρχίσουμε κυρίες και κύριοι, αν θέλετε. Μπορούμε να αρχίσουμε. Κυρίες και κύριοι, ένα θερμό καλώς ήλθατε. Καλωσορίζω ιδιαίτερα στην απογευματινή μας συνεδρίαση στην Ακρόαση τους εμπειρογνώμονες που έχουμε προσκαλέσει, που θα παρουσιάσω ονομαστικά αργότερα, όχι τώρα όμως. Στην Ευρώπη, στον ενεργειακό εφοδιασμό και την ασφάλειά του, πάντα έχει ενδιαφέρον η συζήτηση μετά τη Φουκουσίμα, αφότου για παράδειγμα ένα μεγάλο κράτος μέλος ε, ε, σταμάτησε την πυρηνική ενέργεια και θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις ε, για τις ανανεώσιμες. Η Ομοσπονδιακή Γερμανία και ποιο κόμμα κυρία Μπιούτιχόφερ, θέλετε να τα ακούσετε βλέπω. Η Τσεντεού, το κόμμα μου, η καγκελάριο μου τα αποφάσισε αυτά για να σα καθησυχάσω. Αν καθησυχάζετε, λέω ότι εγώ έχω διαφορετική γνώμη. Δεν πρόκειται όμω περί αυτού σήμερα. Ει ό,τι αφορά το, την ικανότητα αποθεματικών έχουμε πρόβλημα, γιατί η σπάνιση των ενεργειακών πηγών εξελίσσεται και ε, σε πολλά μέτωπα έχουμε δυσκολίες. Το φυσικό αέριο είναι μια ενδιαφέρουσα λύση για τα ορυκτά καύσιμα που έχει το πλεονέκτημα περιορισμένων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης ε, το φυσικό αέριο συνδυάζεται καλά και με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί οι ανανεώσιμες πηγές, ιδιαίτερα ολική και ηλιακή, ε, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το σκέφτονται αυτό ε, πολλά κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν το αέριο. Ξέρουμε ότι 60% του φυσικού αερίου σήμερα εισάγεται από τρίτες χώρες. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχει εξάρτηση 100% από τις εισαγωγές. Όλοι γνωρίζουν ότι η μεγάλη εξαγωγή ε, είναι η Νορβηγία και η Ρωσία αλλά και κάποιες αφρικανικές χώρες. Εμείς ε, ε, έχουμε αυτή την εξάρτηση από τις εισαγωγές που πρέπει να την μειώσουμε και πρέπει να σκεφτούμε άλλες λύσεις. Γι' αυτό εξετάζουμε ως εναλλακτική και το σχισολιθικό αέριο το δυναμικό είναι 216 ε, φορές περισσότερο από το φυσικό αερίο στη Γερμανία. Πολλές τεχνικές πρόοδοι έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια για την εκμετάλλευση και στην Ευρώπη της δυνατότητας αυτής. Είναι εγχώρια πηγή ενέργειας, αλλά υπάρχουν και διάφορες επιφυλάξεις, εμπόδια ε, και η Επιτροπή Περιβάλλοντος μας έκανε μια σχετική ακρόαση. Η συζήτηση δεν γίνεται μόνο εδώ, αλλά και σε πολυάριθμα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε εκείνα τα κράτη-μέλη, τα οποία ε, επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την προβληματική, γιατί έχουν κοιτάσματα σχιστολιθικού αερίου, ε, εκμεταλλεύσιμα, και γι' αυτό ζητήσαμε να κάνουμε μια ακρόαση για να ασχοληθούμε πιο σε μεγαλύτερο βάθος με το θέμα αυτό και έχουμε μία σειρά ειδικών που προσκαλέσαμε, ε, είναι μεγάλος ο αριθμός τους και γι' αυτό θα πρέπει να ε, κάνουμε εξοικονόμηση χρόνου γιατί έχουμε χρόνο μέχρι τις 17 και 30. Καλωσορίζω τον κύριο Μπεσόν, τον κύριο Καραμπούλα, τον, κύριο Βόγαν, τον κύριο Χάουρθ τον κύριο Πίστρο και τον κύριο Ράινικε και νομίζω ότι πρόφερα τα ονόματα σωστά αλλιώς ε, διορθώστε με αργότερα. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο ε, της ε, Διεθνούς Ένωσης Ενέργειας, του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, τον κύριο Κρίς Μπεσόν. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Για να δούμε αν μπορούμε να δούμε τις διαφάνειες. the folder This should be the one that's labeled number one. Yep, that's the one, and put it in. So while this uh, comes up on the screen, now let me... Λοιπόν, σιγά σιγά θα τα δείτε στην οθόνη. Εγώ λέγομαι Chris Besson για να σας συστηθώ στο μεταξύ από τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας. Μου ζητήθηκε να κάνω την εισαγωγή στην ε, ακρόαση αυτή για να σας μιλήσω για τις δυνατότητες που προσφέρει το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Θα σας εκθέσω την άποψη της ε, υπηρεσίας μας μετά την έκθεση την οποία δημοσιεύσαμε για την ενέργεια ε, το Νοέμβριο και θα έχουμε και την έκθεση Golden Age of Gas που θα την ε, έχετε ίσως υπόψη δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο και εκεί εκφράζονται οι προβλέψεις για το σημαντικότερο ρόλο που θα παίξει το φυσικό αυτό αέριο την επόμενη 20 ετία, γιατί αυτό είναι ο χρονικός ορίζοντας που μας απασχολεί, 20 ετία συνήθως. Και επειδή είναι ευκολότερη η παροχή του μη συμβατικού, του αντισυμβατικού και συγκεκριμένα του σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Έχουμε λοιπόν περιγραφή ενός σεναρίου στην έκθεση ε, που δεν είναι βέβαια το πιο πιθανό. Το σενάριο αυτό ε, λέει ότι θα προωθηθεί η χρήση αυτού του φυσικού αερίου μέσω της πολιτικής και άλλων εργαλείων. Εγώ από τις διάφορες εκθέσεις το Energy Outlook, αυτή την έκθεση που σας είπα το Ιουνίου, θα αντλήσω κάποια στοιχεία τα οποία θα σας ε, παρουσιάσω. Πρώτα απ' όλα σε παγκόσμιο παιδί και μετά θα επικεντρωθώ στην Ευρώπη. Άρα ουσιαστικά θα είναι εισαγωγική η ομιλία μου και μετά θα ακολουθήσουν πιο εξειδικευμένες ομιλίες από τους υπόλοιπους του πάνελ. Λοιπόν, βλέπω ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω αυτό το μηχάνημα here? No, to the side. Oh, this one. Okay. So many. This is on off indeed. Wow, wonderful. All right, so let's yeah. try it. Great. Thank you. So as I'm the first speaker, I will. Uh... Είμαι λοιπόν ο πρώτος ομιλητής και θα σας δώσω έναν ε, ορισμό εργασίας ε, για το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Ορισμένοι ομιλητές που θα ακολουθήσουν είναι γεωλόγοι, ίσως uh με διορθώσουν λοιπόν στον ορισμό, αλλά πιστεύω ότι ο ορισμός μου θα είναι η βάση. Είναι ουσιαστικά λοιπόν ε, το φυσικό αυτό αέριο βρίσκεται σε πετρώματα τα οποία εμείς τα ονομάζουμε εν γέννη, σχιστολιθική άνεργο, άργυλο. Ε, Ουσιαστικά πρόκειται για ένα πέτρωμα που είναι πλούσιο σε οργανική ύλη, σε αργύλους, ε, πολύ χαμηλής διαπερατότητας. Αυτό σημαίνει ότι είναι δύσκολο να εξοριχθεί αέριο από αυτό το πέτρωμα και εν γέννη καλύπτει, σε σχέση με το συμβατικό φυσικό αέριο, καλύπτει μεγάλες εκτάσεις. Ε, οι δεξαμενές δηλαδή γεωγραφικά εκτείνονται και είναι και μεγάλο το πάχος επίσης συνήθως των δεξαμενών αυτών. Ίσως το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό είναι ότι μέχρι πριν από μια δεκαετία δεν θεωρείται καθόλου οικονομικά συμφέρουσα η παραγωγή αυτού του φυσικού αερίου. Υπήρχε η παραγωγή των οριζόντιων, μάλλον υπήρχε η χρήση οριζόντιων φρεατίων και τώρα με την υδραυλική ρογμάτωση σε πολλαπλά επίπεδα και στη ΣΥΠΑ είναι η μέθοδος αυτή που χρησιμοποιεί πιο πολύ, έχουν ε, βελτιωθεί οι προοπτικές. Θα σας εξηγήσουν οι συνάδελφοι λεπτομέρειες για την τεχνική αυτή, το hydraulic fracturing, την υδραυλική ρογμάτωση, οπότε εγώ δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες. Ας δούμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ποιες είναι αυτές ε, οι αντισυμβατικές ε, πηγές. Ε, δεν ξέρω αν βλέπετε καλά την οθόνη. Το μπλε είναι τι έχει ήδη παραχθεί, το ήδη ε, παραχθέν φυσικό αέριο. Η κίτρινη και η δεύτερη στήλη είναι το συμβατικό αέριο. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να διαβάσει και να ξεχωρίσει δύο από τα δύο και στη δεξιά στήλη για κάθε μία από τις περιοχές που έχουμε στην οθόνη βλέπουμε το αντισυμβατικό αέριο με το σχιστολιθικό είναι αυτό το μόβ χρώμα και το λεγόμενο συμπαγές χαμηλής διαπερατότητας, tight gas στα αγγλικά, ε, είναι η άλλη, ε, το άλλο χρώμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα Μιλάμε για ανακτήσιμες ε, μη ε, συμβατικές πηγές, πόροι, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Δεν ε, έχει χαρτογραφηθεί πάρα πολύ καλά οι σχιστόλιθοι. Ξέρουμε που βρίσκονται εν γέννη. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μια καλή λίγο πολύ ιδέα για το πόσο φυσικό αέριο περιέχει το πέτρωμα αυτό, αλλά δεν γνωρίζουμε σχεδόν καθόλου πόσο μπορεί να ανακτηθεί ε, πόση η ποσότητά τους. Στις ΕΠΑ αυτή τη στιγμή έχουμε αρκετή εμπειρία για να εκτιμήσουμε αρκετά ε, ικανοποιητικά την ανάκτηση του φυσικού αερίου, αλλά στις περισσότερες άλλες περιπτώσεις ε, προβαίνουμε μόνο και μόνο σε εικασίες. Μιλάμε για πολύ μεγάλες ποσότητες, συνήθως αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας ποιο είναι το ανακτήσιμο κομμάτι. Λοιπόν, να δώσουμε κάποια στοιχεία Με τις νέες τεχνολογίες, το μη συμβατικό αέριο είναι πλέον ε, οικονομικό, είναι, επομένως διπλασιάζεται η δυνατότητα, διπλασιάζεται η ποσότητα φυσικού αέριου μαζί με το συμβατικό. Δεν είναι δηλαδή και τόσο μικρά τα αποθέματα αντισυμβατικού φυσικού αερίου. Βλέπετε τις, ε, ε, τα στοιχεία αυτά στη διαφάνεια. Ουσιαστικά το φυσικό αέριο από τη σχιστολιθική άργυλο διπλασιάζει τα αποθέματα φυσικού αερίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Βλέπουμε ότι υπάρχει διπλασιασμός, παρόλα αυτά στην Ευρώπη είναι μικρές ποσότητες, μικρές ποσότητες ε, των πόρων τέτοιου φυσικού αερίου σε σχέση με άλλες υπήρους. Αυτό το γράφημα σας δείχνει τους ανακτήσιμους πόρους ασχιστολιθικού φυσικού αερίου σε κάποιες ε, χώρες ε, ε, μέλη του ΟΣΑ της Ευρώπης. Λίγες δεν είναι από την Ευρώπη όπως βλέπετε, περισσότερες είναι από την Ευρώπη. Βέβαια δεν είναι ένας πλήρης πίνακας, προέρχεται από μια έκθεση ε, του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας, ε, ERI λέγεται η ε, συμβουλευτική εταιρεία που δημοσίευσε αυτή τη μελέτη και πρόκειται για κάποιες εκτιμήσεις για τους πόρους σχιστολιθικού φυσικού αερίου. Λείπουν κάποιες χώρες όπου γνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημαντικά αποθέματα όπως η Ισπανία, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο γράφημα αυτό παρότι ίσως τα αποθέματά της είναι τόσο μεγάλο όσο κάποιον από τις χώρες που αναφέρονται σε αυτό το γράφημα. Το βασικό επιχείρημα πάντω είναι ότι υπάρχει σχιστολιθικό φυσικό αέριο σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε όπω και σε πολλέ χώρε ε, του κόσμου. Άρα είναι λιγότερο συγκεντρωμένο αν θέλετε από ότι το συμβατικό αέριο που είναι στη Ρωσία κυρίως ε, γενικά στην Πρωτοσοβιετική Ένωση και στη Μέση Ανατολή. Αυτοί, οι χώρε αυτέ έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα συμβατικού φυσικού αερίου, το ίδιο ισχύει και ε, για την Ευρώπη δηλαδή συνολικά τώρα, παγκόσμια, βλέπετε την εικόνα και βλέπετε και την προοπτική των επόμενων 20-25 ετών μέχρι το 2035. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όλο και ε, περισσότερο θα έχουμε αντισυμβατικό φυσικό αέριο. Βλέπετε με το ε, μπλε κάτω είναι το συμβατικό Και όσο περνά ο καιρός βλέπουμε ότι το αντισυμβατικό θα καταλαμβάνει ένα όλο και μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής φυσικού αερίου παγκοσμίω. Όπως ανέφερα, το σχιστολιθικό φυσικό αέριο είναι παρόν σε πολλές χώρες, επομένως ε, περιμένουμε γενικώ ε, το αντισυμβατικό και ειδικώ ε, το σχιστολιθικό φυσικό αέριο να εμφανίσει. να κάνει την εμφάνισή το επόμενα 15-20 χρόνια σε πολλές χώρες εδώ. Δεν βλέπουμε τις ε, ευρωπαϊκές χώρες, γιατί ουσιαστικά είναι μικρό το ποσοστό ε, σε σχέση με άλλες χώρες, αυτές που αναφέρονται συγκεκριμένα εδώ. Αυτά που δεν μπορείτε να τα διαβάσετε μάλλον ε, είναι σε τρεις κυβικών μέτρων. 23 έχει η Ευρώπη, τόσο σε συμβατικό όσο σε μη συμβατικό, ανακτήσιμο φυσικό αέριο και αυτά βέβαια πρέπει να τα συσχετίσετε με μονάδες τις οποίες ίσως γνωρίζετε καλύτερα. Η κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι περίπου 500 δις κυβικά μέτρα το χρόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι 23 είναι 40 χρόνια περίπου. Άρα συμβατικό είναι σημαντικό 80 χρόνια κατανάλωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα Πρέπει να υπάρχουν οι πόροι, πρέπει να υπάρχουν αυτά τα ε, κοιτάσματα σχεστολιθικού φυσικού αέριου, αλλά αυτό που θα περάσει στην μελλοντική παραγωγή ουσιαστικά είναι οι παράγοντες που καταγράφονται, ή τέλο πάντων οι βασικοί παράγοντες, ε, τα οικονομικά, τα ποσοστά, οι συντελεστές ανάκτησης, ε, η ζήτηση, και ρυθμίσεις, κανονισμοί. Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά, και ρυθμισεις κανονισμοι οτι αφορα τα οικονομικα πιστευει ο κόσμος ότι οικονομική τιμή ε, φυσικού αερίου στις ΗΠΑ για την ανάκτηση μη συμπατικού ίσχυση του αληθικού φυσικού αερίου είναι περίπου τη τάξεω των 6 δολαρίων ε, ανά MBTU. Έχω κάνει και τη σχετική μετάφραση γιατί χρησιμοποιούμε εμεί τα κυβικά εκατοστά συνήθω και βλέπετε λοιπόν την αντιστοιχία. Έχουμε ένα συνδυασμό παραγόντων υπάρχει η ανάγκη να έχει κάποιο την άδεια για να μπορεί να παράγει και υπάρχουν και πολλά ρευστά, τα ρευστά υγρά φυσικού αερίου, τα οποία παράγονται και τα οποία μπορούν να πουληθούν ε, στην ε, τιμή του αργού πετρελαιπομένως ε, με την ψηλή τιμή του αργού πετρελαίου τα τελευταία χρόνια είναι οικονομικές οι γεωτρήσεις αυτές που δεν θα ήταν αν παρήγαγαν μόνο φυσικό αέριο. Επομένως πράγματι η οικονομική τιμή ε, θα είναι υψηλότερη στην Ευρώπη σε σχέση με τη ΣΥΠΑ και αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Πρώτα απ' όλα τη δομή της, ε, του κλάδου, της βιομηχανίας που είναι πολύ μικρότερη, το διοκτησιακό καθεστώς των γεών είναι διαφορετικό, περιβαλλοντικές συνθήκες διαφορετικές. Πόσο υψηλότερη τώρα η τιμή δεν το ξέρουμε ακόμη. Κάποιοι συνάδελφοι από τον κλάδο που θα ε, μιλήσουν μετά από μένα ίσως δώσουν, ίσως και δεν δώσουν. αριθμητικά στοιχεία δεν ξέρω αλλά θα το μάθουμε αυτό τους επόμενους 6 με 12 μήνες. Οι πρώτες γεωτρήσεις, ε, οι δοκιμαστικές γεωτρήσεις είναι κατ' ουσίαν στην Πολωνία που είναι πρωτοπόροι στον τομέα αυτό και εκεί πιστεύω θα έχουμε και κάποια επίσημα δεδομένα για τις τιμές που θα χρειαστούν ώστε να είναι οικονομικά αυτά τα φράτη, αυτές οι γεωτρήσεις. Ό,τι αφορά τους συντελεστές ανάκτησης, ουσιαστικά είναι γνωστά τα στοιχεία, βασίζονται και εξαρτώνται από το κοίτασμα ε, του σχιστόλιθου και βλέπουμε και στη ΣΥΠΑ αλλά και εκτός είπα στην Ευρώπη που ε, αρχίζουμε τώρα τις έρευνες, ε, είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που θα καθορίσει και τη ζήτηση που είναι σημαντικός παράγοντας επίσης και περιβάλλον, κανονισμοί, ρυθμίσεις θα σας τα ε, πω στη συνέχεια αλλά θα επανέλθουν με σίγουρος και άλλοι ομιλητές σε αυτά. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για τη ζήτηση. Η περισσότερη ζήτηση, η αύξηση της ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο τα επόμενα 25 χρόνια θα προέλθει κατά πάσα πιθανότητα από τις αναπτυσσόμενες χώρες, Κίνα, Ινδία και ούτω καθεξής. Δεν σας εκπλήσει ιδιαίτερα αυτό. Νομίζω ότι έχει προεξοφληθεί η ζήτηση σε διάφορα σενάρια το 2035 σε σχέση με το 2008. Βλέπουμε παντού αύξηση, αλλά κυρίως και κατά πρώτο λόγο σε αναπτυσσόμενες χώρες. Αυξάνεται όμως σε κάποιο βαθμό και στην Ευρώπη. Στο γράφημα αυτό συγκεκριμένα για την Ευρώπη βλέπετε τα στοιχεία. Με γαλάζιο έχετε την προσδοκόμενη αύξηση στην περίπτωση του χρυσού αιώνα Golden Age ε, που σας είπα ε, Golden Age of Sale και βλέπετε και τις εισαγωγές. Βλέπουμε ότι αυξάνεται και αυτό. Γιατί λοιπόν, παρότι πιστεύουμε ότι θα έχουμε παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου, γιατί έχουμε και αύξηση των εισαγωγών, αυτό το εξηγεί το επόμενο γράφημα που βλέπουμε σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε ένα ε, ανάλογο γράφημα και για την Ευρώπη, αλλά εγώ σας ε, δείχνω τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο για να καταλάβετε τι εννοώ. Ποιο είναι το βασικό θέμα. θα μειωθεί η παραγωγή των, ήδη, ε, γιών που ήδη παράγουν, ε, των περίμετρο από τα οποία μπορούμε να εξορίξουμε ήδη φυσικό αέριο. Αυτό ισχύει και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έχουμε μείωση λοιπόν πάρα πολύ γρήγορη και πολύ από τη δουλειά πρέπει να κάνει, η βιομηχανία έχει να κάνει και με την παραγωγή αερίου αλλά και με την ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση. Και θα πρέπει να αντικατασταθεί η παραγωγή από, τους, ε, από τις φυστάμενες γεωτρήσεις, ε, να ε, βρεθούν δηλαδή υποκατάστατα πετρώματα. Το γαλάζιο, το ανοιχτό εκεί στην Ευρώπη και το λίγο πιο σκούρο είναι κάποια γέες που πρέπει να αναπτυχθούν και δεν έχουν ακόμη ίσως και βρεθεί. Είναι μικρότερο το κομμάτι αυτό γιατί η Ευρώπη κυρίως παράγει συμβατικό αέριο και σε σχέση με το αντισυμβατικό που βλέπετε πάνω-πάνω είναι ανάλογη εικόνα στην Ευρώπη όπως και για την υφήλιο εν γέννη. Θα αυξηθούν λοιπόν με ταχύς ρυθμούς ε, το σχιστολιθικό και το ε, ε, μη συμβατικό, αλλά θα πρέπει να αντισταθμιστεί η μείωση της παραγωγής του συμβατικού αερίου και γι' αυτό, επειδή αυτό θα είναι δύσκολο, θα, έχει μεγάλο ρόλο πάλι, ε, θα έχουν μεγάλο ρόλο οι εισαγωγέ που θα αυξηθούν και αυτές. Περιβαλλοντικές τώρα πτυχές. Έχει γίνει πολλή συζήτηση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, φαντάζομαι έχετε διαβάσει. Υπάρχουν ανησυχίες περιβαλλοντικές σε σχέση με το συμβατικό αέριο και συγκεκριμένα με την τεχνική που χρησιμοποιείται για την παραγωγή αερίου, αυτά τα οριζόντια, αφράτη, οριζόντιες ε, ε, γεωτρήσεις ε, με την πολυεπίπεδε, με τις πολυεπίπεδες ρηγματώσεις, υδραυλικές ρηγματώσεις. Επίσης πρέπει να δούμε τι γίνεται με το νερό το οποίο παράγεται, με τις, εκπομπέ με αερίων, τη χρήση της γης, γιατί ε, ξέρουμε ότι στην ε, ε, εξόριξη του φυσικού αερίου χρειάζεται, χρειάζονται πολλά φρέατρα, πολλές γεωτρήσεις και επομένως υπάρχει και ζήτημα και με τον υδροφορίζοντα και στη ΣΥΠΑ έχει προκύψει αυτό. Όταν έχουμε λοιπόν κάποιες βέλτιστες πρακτικές βιομηχανικές και ρυθμιστικές, αυτές οι ανησυχίες υπερβαλλοντικές πιστεύω ότι μπορούν να μετριαστούν. Δεν έχει συμβεί πάντοτε αυτό βέβαια στη ΣΥΠΑ και φαντάζομαι το ίδιο θα ισχύσει και στην Ευρώπη. Αλλά αν χρησιμοποιούνται ε, καλές πρακτικές, εδώ βλέπετε τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα από φυσικό αέρα σχιστολιθική άργυλο. Βλέπετε εδώ για τη χρήση σε μία κάμινο, σε ένα ε, εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας. πάνω χάρη, ε, αριστερά βλέπετε για το συμβατικό, δεξιά με το σχιστολιθικό αέριο, χωρίς βέλτιστες πρακτικές. Με τις βελτιστές ε, πρακτικές βλέπετε ότι είναι μικρή η διαφορά, ε, αλλά αν δεν είναι κανείς προσεκτικός μπορεί να έχει σημαντικές ε, αποκλήσεις και διαφορές και κυρίως με την εξαέρωση του αερίου. Θα ήθελα τώρα κοντεύω να τελειώσω την παρουσίασή μου, αν και μακρηγόρησα λίγο και στο συγγνώμη γι' αυτό. Λοιπόν, οι εκπομπέ δεξιδίου του άνθρακα, ε, γενικά για τη βιομηχανία φυσικού αερίου, πολλοί μιλούν ε, για το αέριο παρουσιάζοντα το στη λύση για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Η μελέτη μα δείχνει ότι αυτό δεν ισχύει απόλυτα. Εγώ σα δείχνω τη διαφορά μεταξύ αυτού του τυπικού σεναρίου ε, και του σεναρίου Golden Age of Gas όπου φτάνουμε στα άκρα λίγο με τις υποθέσεις μας ε, και βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση ε, διοξιδίου του άνθρακα γιατί έχουμε μικρότερη πυρηνική ενέργεια και λιγότερες ΑΠΕ, ανανεώσιμες πηγές, πολύ λιγότερος άνθρακας όμως οπότε υπάρχει ένα αντιστάθμισμα αλλά το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι δεν υπάρχει ε, και τόσο μεγάλο κέρδος σε ό,τι αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα αν προσπαθήσουμε να φτάσουμε στα άκρα με τη χρήση του φυσικού αερίου. Σε κάποιες εβδομάδες από τώρα ε, θα έχουμε ε, το World Energy Outlook ε, του χρόνου αυτού, τον Νοέμβριο συγκεκριμένα, και θα έχουμε και κάποια ενημερωμένα, επικαιροποιημένα στοιχεία για το φυσικό αέριο και τους πόρους φυσικού αερίου και ίσως και κάποια από τα αποτελέσματα τα οποία θα μας δώσουν οι Πολωνοί άλφοι με τις πρώτες τους γεωτρήσεις στην Πολωνία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ähm, Ευχαριστούμε πολύ για τα στοιχεία αυτά κύριε Μπεσόν. Χωρίς διάλειμμα προχωρούμε στον επόμενο γύρο όπου θα μιλήσουμε για βιομηχανικά θέματα εμπορικά, ε, οικονομικά. Ο κύριος ε, Καραμπούλα είναι αντιπρόεδρος της Oil and Mining PGNIG, ε, πολωνική εταιρεία πετρελαίου και αερίου. Προσέξτε, έχουμε πολλούς ομιλητές προσκεκλημένους, πρέπει εμείς να είμαστε σύντομοι. Εγώ θέλω να μπω στον κατάλογο για αργότερα. Εντάξει, πρώτος θα είστε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μπορούσα, μπόρεσα στις 27 Ιουνίου να δω κάποιους από εσά στην Πολωνία. Χαίρομαι που επανέρχομαι και να κάνω μια παρουσίαση για την εταιρεία ε, αυτή στην Πολωνία και τις εξελίξεις του στο σχιστολιθικό. Εμείς είμαστε πλήρως ολοκληρωμένη εταιρεία στον τομέα της ε, εξόρυξης. Ε, επίσης είμαστε με τη Gazprom και κάνουμε και, στην, και αποθήκευση και κάνουμε διαχωρισμό unbundling είναι διαφορετική η εταιρεία στην Πολωνία η οποία είναι η ιδιοκτήτρια και διαχειρίζεται τα συστήματα υψηλής μετάδοσης. Επίσης ε, ε, συμμετέχουμε στην ε, διανομή και στο λιανεμπόριο. Έξι εκατομμύρια πολωνικές οικογένειες εφοδιάζονται. Κάποιοι μας θεωρούν εθνική εταιρεία, 72% και παραπάνω ε, το έχει το κράτος, το υπόλοιπο είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο της Βαρσοβίας, η κεφαλαιοποίηση τώρα είναι περίπου 9 δις δολάρια. Σήμερα όμως ε, θέλω να σας κάνω κάποια σχόλια σχετικά με την ε, οικονομική βιωσιμο... εμπορική βιωσιμότητα της εταιρείας. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια για την εταιρεία μας σχιστολιθικού αερίου. Ε, έχουν ήδη ε, αναφερθεί ε, πολλές δυνατότητες για την εμπορική βιωσιμότητα. Δεν θα μιλήσω μόνο για την οικονομική σκοπιμότητα των έργων ή για την κερδοφορία του σχιστολιθικού αερίου. Ε, αυτό θα είναι το τελευταίο. Αλλά θα αρχίσω ε, με κάποια θέματα περιβαλλοντικά. Και αυτό που είναι πραγματικά σημαντικό είναι όχι μόνο να πούμε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα που τα ξέρουμε κι εμείς, αλλά είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσουμε με το σωστό τρόπο με την κοινή γνώμη. Και αυτό που κάναμε για να κατανοήσουν και άνθρωποι που δεν τα γνωρίζουν είναι ναι, κάνουμε μικρές σχισμές, κάνουμε ρογμάτωση. Τον Ιούλιο του 2010 κάναμε ε, το πρώτο, την πρώτη υδρορογμάτωση στην Πολωνία και δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν ήταν πολύ επιτυχή. Δεν παραιτηθήκαμε όμως. 18 Σεπτεμβρίου του 2011 στο Λούμποτζιν είχαμε επιτυχία μετά από ε, ε, μια αργμάτωση ε, σε κατακόρυφο φρεάτιο μπορέσαμε να βγάλουμε αέριο. Αργότερα θα επανέλθω σε αυτό. Μια άλλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Πολωνία είναι η Freetex Resources. και είχαν και εκείνη επιτυχία έκαναν επίσης γεώτρηση, κατακόρυφη και έκαναν πολλαπλή ρογμάτωση στο οριζόντιο φρεάτιο. Τι έχουμε μέχρι τώρα στην Πολωνία. Έχουμε 10 φρεάτια ε, γεωτρήσεις για το συστολιθικό αέριο αποκλειστικά και 3 φρεάτια ε, όταν ε, έγινε η διαδικασία της ρογμάτωσης. Όμως για να πάμε τώρα στην εμπορική βιωσιμότητα και σε αξιόπιστες πληροφορίες, τι κάνουμε εμείς ως εταιρεία Picnic. Ε, έχουμε επαφή με τις τοπικές κοινότητες, συμμετέχουμε σε διασκέψεις, σε συνέδρια, μιλούμε στον ντόπιο πληθυσμό, στα δημοτικά συμβούλια, ε, μιλάμε με τους αγρότες ε, που αγοράζουμε ή μισθώνουμε γη από τους αγρότες για να κάνουμε τη δουλειά μας. Και όταν συναντούμε αυτούς τους ανθρώπους και εξηγούμε πολλά θέματα, βλέπουμε αν γιατί πολλές πληροφορίες δίνουμε για την ε, υδρορογμάτωση. Κάποιοι έχουν ερωτήσεις, αλλά και εμείς είμαστε ε, πάρα πολύ ευτυχείς να απαντήσουμε και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την τελευταία φορά που σας συνήντησα στις 27 Ιουνίου τρέχοντος, ε, οργάνωσα συναντήσεις στο Μάρκο Βόλα και αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι επανήλθαμε ένα χρόνο μετά την υδρορογμάτωση στην τοπική κοινότητα για να δείξουμε πώς ε, ε, φέραμε στην ίδια κατάσταση που ήταν η γη πριν κάνουμε την εξόρυξη Είπαμε ότι θα επανέλθουμε. Τους το εξηγήσαμε. Θα ξαναγυρίσουμε στις διάφορες περιοχές της Πολωνίας. Ε, στις 7 και 9 Σεπτεμβρίου κάναμε στην Κρινίτσα άλλη συνάντηση όπου δείξαμε σε, στο ευρύ κοινό διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για τις γεωτρήσεις και, γιατί, και εργαλεία αργωμάτωσης. Επίσης κάναμε στις 27 Σεπτεμβρίου μια άλλη συνάντηση στο Λουμπάτσι Νόβα για να δείξουμε πάλι στην τοπική κοινότητα τι πρόκειται να κάνουμε τους επόμενους μήνες όταν θα προχωρήσουμε ε, σε οριζόντια γεώτρηση και πολλαπλή ρογμάτωση. Ε, στην Πολωνία όταν τέθη το ερώτημα να παράγουμε ή να μην παράγουμε συστολιθικό αέριο, η απάντηση είχε ως εξής. Γενικά, 73% των Πολωνών είναι υπέρ της παραγωγής του αερίου αυτού του σχιστολιθικού, shale gas. Όμως πάντα υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά την παραγωγή στην πίσω αυλή μου. Γιατί σε πολλές χώρες της Ευρώπης θα δείτε ανθρώπους να λένε όχι, δεν θέλω στην πίσω αυλή μου. Στην Πολωνία πάνω από το 56% λένε ναι, δεν έχω αντίρρηση στην παραγωγή και αξιοποίηση του αερίου στην πίσω αυλή μου, σε ε, γη που μου ανήκει. Αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας. Για να ξαναγυρίσουμε στην εμπορική βιωσιμότητα, ένα άλλο θέμα που πρέπει να θέσουμε αφορά την τεχνολογία και τη γεωτεχνική κατανόηση του θέματος. Ε, στους δύο αυτούς τομείς μπορούμε να πούμε ένα πράγμα. Πρώτον, εμεί ω εταιρεία Peganica χρησιμοποιούμε την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία. Ε, όλες οι διαδικασίες ρογμάτωσης γίνονται με τη βοήθεια και την στήριξη της Χάλι Μπάρτον. Το 2010, πριν από ένα χρόνο και πριν από ένα μήνα τώρα, η Χάλι Μπάρτον, ε, μια ομάδα από τη Γερμανία, ήρθε στην Πολωνία και έκανε την ε, υδρορογμάτωση. Ε, μπορώ να σας περιγράψω λεπτομερώς πώς γίνεται αυτό. Τώρα θα πω ένα πράγμα. Χρησιμοποιούμε 1.600 κυβικά μέτρα νερού, αντλούμε σε ένα φρεάτιο 3.000 μέτρα βάθος. Και η δουλειά αυτή ε, κράτησε 210 λεπτά. Όλα έγιναν σύμφωνα με, το, με τα σχέδια και τις βέλτιστες διαθέσιμες πρακτικές. Δεν υπήρξε ε, καμία περιβαλλοντική επιπλοκή και κάτι ακόμα. Η δουλειά ρογμάτωσης που κάναμε στη Μαρκοβόλα πριν από ένα χρόνο παρακολουθήθηκε από το Πολωνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έκαναν κάτι που συνήθως δεν γίνεται κατά ανάγκη, αλλά επειδή ήθελαν να τσεκάρουν και να επαληθεύσουν ότι όλα είναι εντάξει, και ότι ό,τι κάναμε είναι αυτό που έπρεπε να κάνουμε, ήρθαν και έκαναν έλεγχο. Ε, το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν ξεκάθαρο. Είπαν ότι κάναμε τα πάντα νομοτύπως και να πούμε και κάτι ακόμα. Στην Πολωνία έχουμε 130 ε, νόμους και άλλες νομοθεσίες που ρυθμίζουν την εξόριξη και παραγωγή αερίου. Ε, ε, ε υποκείμεθα στο mining law το νόμο για τις εξορίξεις ε, που διαφέρει από την, τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά ακόμα. Υπογραμμίζω όμως ότι ε, μας έγινε έλεγχος και ε, το αποτέλεσμα είναι ότι συμμορφωθήκαμε σε όλους τους κανόνες, νόμους, κανονισμούς. δηλαδή τα 130 νομοθετήματα τα τηρήσαμε. Κάτι άλλο που πρέπει να πούμε και που κάνει βιώσιμο είναι κάποια θέματα σχεδιασμού και βιομηχανικές εφαρμογές. Δύο σχόλια πρέπει να κάνουμε εδώ. Το ένα είναι η, τεχνολογία της υδρορογμάτωσης που είναι κλεπτισμένη, ε, είναι ιδιαίτερα υψηλές οι πιέσεις, ε, οι 360 μπαρ, οι ε, ατμόσφαιρες στο νερό, αλλά εμείς έχουμε τέτοιες, τις ξέρουμε στην Πολωνία αυτές, παράγεται ήλιο. Μία χώρα στην Ευρώπη, η Πολωνία, ε, στο, το δικό μας ε, εργοστάσιο παράγει ήλιο στο Χοντολάνοφ ε, και δουλεύουμε σε πολύ χαμηλές, ακραία χαμηλές θερμοκρασίες. Αν κάποιος έχει αμφιβολίες για το αν μπορούμε να διαχειριστούμε την υδρορογμάτωση, η απάντηση είναι ναι και πάλι ναι πάνω από 30 χρόνια δουλεύουμε σε ακραία χαμηλές θερμοκρασίες και είμαστε σημαντικοί παράγοντες σε ό,τι αφορά το ήλιο. Δεν θα μιλήσω για διάφορες χρήσεις του ηλίου στον κόσμο. Εφτά χώρες μόνο όμως μπορούν να πούν ότι παράγουν ήλιο. Η Πολωνία είναι μία από αυτές. Ε, ένα άλλο σημαντικό θέμα. Ε, η συνεργασία μας με τα πανεπιστήμια. Εμείς ε, έχουμε κάνει το πρώτο βήμα και δημιουργήσαμε ένα κονσόρτσιουμ με Πολυτεχνία της Κρακοβίας, τη IGH, ε, από τα πρώτα, επίσης με την Τεχνολογική Ακαδημία και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Κρακοβίας για το πετρέλαιο. Τεχνολογία πετρελαίου. Θέλουμε να αναπτυχθούμε να εξελιχθούμε, να μάθουμε περισσότερα και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα συμμετάσχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα εντάσει και άλλες χώρες της Ευρώπης. Και το πρόγραμμα αυτό, το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα, βέβαια είναι, γίνεται χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάτι ακόμα ε, σε σχέση με τις υπηρεσίες. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν πολλές γεωτρήσεις τώρα στην Ευρώπη. Αλλά καναδικές εταιρείες, Γένσαν ε, μία από αυτές, ήδη είπε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ να αρχίσει η παραγωγή στην Πολωνία. Επίσης, ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα που αφορά την βιωσιμότητα, τα οικονομικά θέματα. Τα οικονομικά θέματα είναι πολύ σημαντικά. Για να δούμε κάποια νούμερα. Καταρχήν, Ήδη αναφέρθηκε ότι το σχιστολιθικό αέριο ε, οδήγησε σε αλλαγές στη ΣΥΠΑ. Βλέπετε εδώ, ε, ιδιαίτερα βλέπετε την πράσινη γραμμή. Ε, εδώ η τιμή του εισαγωμένου στη ΣΥΠΑ LNG έχουν πάνω από 500 δις κυβικά ε, μέτρα, αλλά εισάγουν και πολύ LNG. Και κάποια στιγμή η τιμή του LNG έφτασε στα 12 δολάρια, ε, μπορεί και 14 και είπαν όχι. Δεν πρόκειται να το δεχτούμε. Εμείς είμαστε πλούσια χώρα, αλλά δεν πρόκειται να δεχτούμε να πληρώνουμε 12 ε, και 14 δολάρια ανά εκατομμύριο BTU. Και άρχισαν να πολλούν και με το συστολιστικό αέριο έπεσε η τιμή. Ήδη είπε ο συνάδελφος ότι υπάρχει τώρα 6 ε, δολάρια ε, και έχουμε φτάσει και στην τιμή των 4,70. Όμως τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αντιμετωπίζουν πια ε, το, τις εισαγωγές της πολύ ακριβές του LNG. δείτε την πορτοκαλή γραμμή, η Ιαπωνία είναι αυτή. Ε, δεν θα πω για την Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία βλέπετε την μείωση στις τιμές LNG, αλλά αυτή ήταν μόνο προσωρινή μετά την κρίση του 2008 και 2009 διότι βέβαια πρέπει να αναφέρομαι ορισμένα πράγματα σχετικά με το τι θα γίνει μετά τη Φουκουσίμα και μετά τις, ε, τους σεισμούς. Για να δούμε τώρα το, διάγραμμα, το γράφημα για την Gazprom. Ε, Όταν μιλάμε για εμπορική βιωσιμότητα πρέπει να μιλήσουμε για τιμές. Βλέπετε εδώ κάποια στοιχεία. Βλέπετε εδώ την κάθετη στήλη γραμμή που είναι η 11η Μαρτίου. Στις 11 Μαρτίου ε, έγινε ο σεισμός, σεισμή μέχρι τις 13. Δύο μέρες κατά στην Ιαπωνία. Και τι έγινε με την πράσινη πράσινη γραμμή η τιμή LNG που ήταν 10 δολάρια ανά 1 εκατομμύριο BTU ανέβηκε στα 16 δολάρια μέσα σε μια μέρα μόνο. Και τι γίνεται στο, στο γράφημα. Βλέπουμε εδώ 15 Μαρτίου μερικές μέρες μόνο μετά τους σεισμούς και πάνω στη βάση των μακροπρόθεσμων συμβολέων, συμβάσεων ε, κανονικά ανεμένετο να πέσει η τιμή. Θα σας δείξω, δυστυχώ δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Εδώ στο γράφημα βλέπουμε επίση την ανάπτυξη, την εξέλιξη τιμών στο άμεσο μέλλον μέχρι το 2014. Παρακολουθούμε τις τιμές χάρη στην ISIS. Αλλά δυστυχώς ε, δεν έχουμε προγνωστικά για μετά το 2014. Ακόμα όμως εδώ βλέπουμε ότι στη γερμανική αγορά οι τιμές θα είναι σε επίπεδα άνω των 12 δολαρίων ανά εκατομμύριο BTU και στο Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι περίπου 10. Και ε, στο, στις Ηνωμένε Πολιτείε, ε, στο Henry Cup, στο Trading Point εκεί, που δεν είναι εικονικό μόνο, γίνεται, γίνονται και παραδόσεις εκεί, ε, χτυπάει μόνο 6 δολάρια. Η διαφορά λοιπόν μεταξύ ΙΠΑ και Ευρώπης είναι διπλάσια, 6 έναντι 12. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας κάνει να σκεφτούμε το σχιστολιθικό πολύ σοβαρά, γιατί αυτές οι εξελίξεις τιμών δεν πραγματοποιούνταν πριν. Παλιά ήταν σε άλλες τιμές το σχιστολιθικό αέριο. Για να ξαναγυρίσουμε για ένα λεπτό στην Ιαπωνία. Όπως ανέφερα, ακόμα ε, το πριν από το Μάρτιο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, οι τιμές για την Ιαπωνία και την Ευρώπη ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Japan Korean Market, ε, στην Ιαπωνική Κορεατική, άρχισε στα 10 δολάρια. Τώρα, έχουμε από τη Mitsubishi Corporation που ξέρουν και ε, είναι εμπορεύονται το LNG, 21 Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι η τιμή χτύπησε τα 16 δολάρια ανά εκατομμύριο BTU. Αλλά ποια είναι η τιμή σήμερα. Η τιμή είναι 17,5 17,5 ε, δολάρια ανά εκατομμύριο BTU. Έξι, μέσα σε 6 μήνες άλλαξε άρδινη η κατάσταση. Και το ερώτημα είναι, έχουμε την πολυτέλεια να πληρώνουμε τέτοιες τιμέ. Η Ιαπωνία μπορεί, πλούσια χώρα είναι. Η Πολωνία όμως δεν μπορεί, γιατί εμεί δεν είμαστε πλούσιοι, όχι ακόμα. Ε, όμως έχουμε τον τρόπο να βελτιωθούμε κατά τη. Τώρα, μιλάμε για τιμέ. Τιμέ εντάξει, αλλά δεν αρκεί να μιλάμε για αυτό. Χρειάζεται να μιλήσουμε και για τη ζήτηση. Υπάρχει μεγάλο κενό. Τι πρόκειται να συμβεί. Θα αυξηθεί η ζήτηση για αέριο, γιατί αυξάνεται η ζήτηση για την ενέργεια στην Ευρώπη. Εμείς πώς θα ανταποκριθούμε στις ανάγκες αυτές το 2030. Σίγουρα το σχιστολιθικό αέριο δεν θα αποτελέσει τη μόνη λύση. Αλλά ας του δώσουμε μια ευκαιρία του σχιστολιθικού αερίου ε, που είναι πλούσιο, πλούσιο σπόρος εδώ στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Πολωνία. Έχουμε στοιχεία από την Πολωνία βέβαια, έχουμε δει και τα, τις σπόρους που υπάρχουν στην Γαλλία, αλλά τις τελευταίες εβδομάδες και το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι έχουν ακόμα μεγαλύτερα κοιτάσματα χάρη στην Κουαντρίλα, μεγαλύτερα από την ε, Πολωνία ας δώσει μια ευκαιρία στο σχιστολιθικό αέριο. Ας δούμε κάποιες αναλύσεις τώρα. Ιδιαίτερα εδώ και πάλι, εδώ, η Σεύρον, με βάση τη Μακένζη, την ανάλυση Μακένζη που δείχνει την τιμή. Τι θα στοιχήσει, ας πούμε, η ανάπτυξη στην Πολωνία. 8, λίγο παραπάνω δολάρια και ο όγκος μπορεί να είναι 40 δις κυβικά μέτρα. Ίσως όλη η Ευρώπη θα μπορεί να πάει στα 240 κυβικά μέτρα το 2020 όλοι μαζί στην Ευρώπη. Δεν ανταγωνιζόμεθα με τη Ρωσία, δεν ε, ε, ανταγωνιζόμαστε την Gazprom, ε, ούτε δεν δίνουμε μάχη με ανεμόμυλους, ούτε με την ηλιακή. Εμείς έχουμε πολλά να κάνουμε ως εταιρείε αερίου. Και άλλοι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Τέλος, ένα θέμα πολιτικό. Εδώ, γιατί ε, ε, τελειώνει και ο χρόνος με εμείς στην Πολωνία, ως εταιρεία Πιντενίκα, αρχίσαμε μια μικρή εκστρατεία. Μην σβήσουμε τη φλόγα της ελπίδας. 100, μέσα σε 140 ώρες, δηλαδή αρχίσαμε την περασμένη Τετάρτη την ε, εκστρατεία. Συλλέξαμε πάνω από 16.000 16 ψήφους Πολωνών που παρακαλούν να μην γίνει κάποια ε, ε, μην αναλυθεί η δράση που θα σταματήσει την εξόριξη Χιστολιθικού αερίου στην Πολωνία. Ε, κάποια νούμερα οικονομικά, εδώ μιλάμε για την τελευταία έκθεση ενός, της Barnet Shale, που είναι από τις πιο αναγνωρισμένες και παλιότερες περιοχές σχιστολιθικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. 9-3 κυβικά πόδια δίνουν περίπου 100.000 θέσεις εργασίας, υπάρχουν στοιχεία οικονομικά. Αλλά επειδή δεν έχω χρόνο, θα... δεν θα τα πω. Τώρα, οικονομικές, δημοσιονομικές επιπτώσεις, πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Αν δούμε το 2030, ας πούμε, και ως Ευρώπη θα εισάγουμε περίπου 280 ε, περίπου εκατομμύρια κυβικά μέτρα αερίου και αν έχουμε 10 δολάρια ας πούμε τιμή ανά εκατομμύριο BTU θα δαπανίσουμε περίπου 98 δις δολάρια. Εμείς πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για να το πούμε διαφορετικά. Η Πολωνία σήμερα εισάγει 10 δις ε, κυβικά μέτρα το χρόνο με αυτή τη τιμή, 10 δολάρια ένα εκατομμύριο BTU, κάθε χρόνο αυτό σημαίνει ότι πανούμε και βγάζουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω από τη χώρα μας 3,5 δις δολάρια. Φεύγουν από τη χώρα μας. Αυτό μπορεί να αλλάξει. Πιστεύω λοιπόν ότι το σχιστολιθικό αέριο θα ωφελήσει την Ευρώπη. Βέβαια πρόκειται να βελτιώσουμε το κλίμα και σίγουρα αυτό ταιριάζει ε, στο σύστημά μας, θα, χρησιμοποιήσουμε, ε, θα, έχουμε ενεργειακή ασφάλεια και εξασφάλιση θέσεων εργασίας. Ένα θα σας πω, ας δώσουμε στον εαυτό μας μία ευκαιρία για να τα καταφέρουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κατευθείαν στο, το λόγο στον κύριο Βόγαν, ε, ο οποίος ε, είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο, από το Καντρίλα Resources, ε, Chief Operating Officer. Να έχουμε υπόψη μας τον χρόνο, γιατί ο τελευταίος ομιλητής δεν θα προλάβει να μιλήσει. Έχετε το λόγο. I'm Eric Vaughn, I'm the Chief Operations Officer of Quadrilla Resources. Γεια σας. Λέγομαι Eric θα σας ε, μιλήσω για την Quadrilla, την εταιρεία που εκπροσωπώ. Να δούμε μετά ποια είναι αυτά τα οποία κάποιοι κλαμβάνουν σε εμπόριο στην ανάπτυξη και ποιος είναι ο οικονομικός αντίκτυπος της ανάπτυξης. Quadrilla Resources λοιπόν είναι μια εταιρεία με βάση το Ενωμένο Βασίλειο στο Lichtfield, στο Staffordshire. Συστηθήκαμε, είμαστε μια ιδιωτική εταιρεία το 2007 ε, μέχρι στιγμής έχουμε δύο γεωτρήσεις και ε, ανοίγουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο Τώρα το τρίτο φρεάτιο, η έκτασή μας που έχουμε άδει είναι 6.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είμαστε ενοποιημένη εταιρεία, δηλαδή έχουμε τις δικές μας υπηρεσίες γεώτρησης, ρογμάτωσης και δοκιμής. Τι θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι είναι φραγμή στην ανάπτυξη, όπως αναφέρθηκαν και κατοπερθώνισμένοι, έλλειψη εξοπλισμού, η πυκνά του πληθυσμού που είναι διαφορετική στη Βόρεια Αμερική, υπάρχει η αντίληψη εκεί ότι αυτή η τεχνολογία, ιδίω η ρογμάτωση που είναι μια νέα τεχνολογία που δεν έχει δοκιμαστεί, πρέπει να γίνουν μελέτε επιπτώσεων και επειδή ε, υπάρχουν και ζητήματα εμπιστοσύνη τη κοινή γνώμη, ε, θα δείτε και στην έκθεση ότι λένε ότι μπορεί να μην υπάρχει αρκετό αέριο, άρα υπάρχει πρόβλημα για την εγγύηση της ανάπτυξης. Αυτό δεν είναι αρκετό. Λοιπόν, το, όπως σας είπα, έχουμε ε, τους δικούς μας ε, στόλους, τα δικά μας ε, φρεάτια, τις δικές μας εξέδρες. είχαμε και μία... ένα γεωτρύπανο που κατασκευάστηκε στον Καναδά και γενικώ καταφέρνουμε οικονομικά να είμαστε σε χαμηλά επίπεδα, δεν χρειαζόμαστε πολλούς προμηθευτέ και μπορούμε να προγραμματίσουμε και τις εργασίες μας όπω αυτό μας εξυπηρετεί καλύτερα. Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία. Αν δείτε τους διάφορους αυτούς, ε, τα διάφορα εργοτάξια, είδαμε ότι ξεκίνησαν να συνεργάζονται με εταιρείε πολύ μεγάλες, γεωτρήσεων και έτσι θα έχουν πολύ γρήγορα τον εξοπλισμό Υπάρχει ήδη ε, πολύ εξοπλισμό και για υδρορογμάτωση που θα είναι έτοιμο και θα έρθει στη, σύντομα στην Ευρώπη. Βλέπετε εδώ την, ε, τα 30 μέτρα ύψους αυτού του, αυτής της ε, διάταξης και μετά βλέπετε και τον εξοπλισμό υδρορογμάτωσης. Βλέπετε τις δεξαμενές νερού αριστερά ψηλά είναι λίγο διαφορετικό όταν γίνεται δρορογμάτωση ε, στην Ευρώπη. Δεν υπάρχουν ε, ε, στην Βόρεια Αμερική ανοιχτά ανοιχτές δεξαμενές. Βλέπετε τις αντλίες τώρα κάτω, τις αντλίες ρογμάτωσης. 15.000 είναι υποδύναμη και βέβαια η δεξιά κάτω πλευρά βλέπετε το φρέα και την κεφαλή του. Ένα άλλο θέμα είναι η δημογραφική πυκνότητα που επίσης είναι διαφορετικά τα πράγματα στη ΣΥΠΑ, τη Βόρεια Αμερική από την Ευρώπη, που μπαίνουμε λοιπόν όλα αυτά τα φρεάτια. έχουμε τις διάφορες ε, εταιρείε. Συνήθως οι εργασίες γίνονται επί τόπου. Τα φρεάτια είναι λιγότερο από 30 μέτρα. και γενικώ προσέχουμε να ε, μην δημιουργούμε και προβλήματα ηχορύπανσης. Έχουμε τα 250 μέτρα, προσπαθούμε να τηρούμε αυτή την απέτηση και δεν χρειάζεται να έχουμε και επιπλέον ηχομονωτικά τυχώματα. Εδώ βλέπετε την, ε, ένα από τα πρώτα φρεάτια, μία από τις πρώτες γεωτρήσεις ε, στο Ενωμένο Βασίλειο. Βλέπετε ότι εκεί δεν έχουμε θέματα με την πληθυσμιακή πυκνότητα. Εδώ βλέπετε πώς ε, θα μπορούσε να δείχνει η Ευρώπη σε λίγα χρόνια αν ξεκινήσει η ανάπτυξη. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν πρόκειται αυτό να πλησιάζει στην ε, πραγματική εικόνα. Ακόμη και αν μπορούσε κανείς να κάνει γεωτρήσεις τέτοιου είδους στην Ευρώπη, αυτό δεν θα ήταν οικονομικά αποδοτικό για τις ε, κατασκευαστικές εταιρείε, γιατί είναι 500.000 ευρώ η όλη επένδυση για τη γεώτρηση όταν χρειάζεται να είναι πολλαπλά τα φρεάτια. Εδώ βλέπετε κάτι ανάλογα με αυτό που γίνεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, δεν μπορώ να σας δείξω βέβαια ακριβώς ε, τις... Ε, δεν, μπορείτε, δεν μπορείτε να δείτε ακριβώς που εργαζόμαστε, αλλά τέλος πάντων κάπου στο μέσο είναι. Πάνω αριστερά κοντά στο ποτάμι εκεί πέρα υπάρχει αυτό το κέντρο και το και εκεί που βλέπετε το ε και εκεί υπάρχει ένα well pad Και εκεί στο τετράγωνο που βλέπετε και εκεί έχουμε ένα well pad, τρία χιλιόμετρα έχει το ένα από το άλλο, αρκετά κοντά στην περίπτωση αυτή. Αν έχετε οριζόντιες 2-3 μπορεί με απόστασή τους να είναι μεγαλύτερη. Επίσης, ε, η τεχνολογία fracturing της αρωμάτωσης θεωρείται ως μια νέα τεχνολογία που δεν έχει δοκιμαστεί. Όμως τα τελευταία 60 χρόνια πάνω από ένα εκατομμύριο φρεάτια χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή και γίνεται και στις, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία, ε, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 80 εξ όσων γνωρίζω χρησιμοποιεί την τεχνική αυτή. Σίγουρα είναι διαφορετική η τεχνική της ρογμάτωσης ε, κατά το παρελθόν σε σχέση με σήμερα. Ε, εντάξει, στη δεκαετία του 80 και του 90 ε, η τεχνολογία είναι αυτή που ακολουθείται σήμερα και στα περισσότερα σιλό. Το EPA έχει κάνει μια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Grand Water Protection Council εξετάζει το θέμα της ε, ε, ρηγμάτωσης και επίσης η Interstate Oil and Gas Compact Commission εξετάζει και αυτή τη διαδικασία και γενικώ έχει εγκριθεί από αυτούς τους αρμόδιους οργανισμούς. Εδώ βλέπετε αριστερά ένα από τα πρώτα ε, εργοτάξια υδρορογμάτωσης, κάτι αντίστοιχο με αυτά που γίνονται σήμερα στην ε, περίπτωση εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού και κάτω βλέπετε ένα άλλο ε, εργοτάξιό μας μία από τις μεγαλύτερες, ε, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που ανέλαβα εγώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, συγκεκριμένα το 1992, που επίσης είχαμε την τεχνική της υδρογραμμάτης με ζελατονοποιημένο νερό. Άρα υπάρχει αυτή η τεχνική εδώ και αρκετά χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα τον ε, περιβαλλοντικό αντίκτυπο, στην Ευρώπη σίγουρα γίνονται κάπως διαφορετικά τα πράγματα σε σχέση με τη Βορεια Αμερική. Ε, σε ό,τι αφορά την έκταση έχουμε κάποια ε, ησυχίες σε σχέση με διαρροές που θα μπορούσαν να μολύνουν τα νερά τα ύδατα, αλλά εμείς έχουμε κάποιες διαπερατές ε, μεμβράνες ε, στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή σε άλλες περιπτώσεις όπως στην Ολλανδία υπάρχει σφράγιση, τοποθετείται ένα ε, προστατευτικό στρώμα, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση διαρροής. Και κάτι άλλο το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ότι έχουμε συνεχή παρακολούθηση του εδάφους ε, για να μην υπάρξει πουθενά κοντά ε, στο εργοτάξιό μας διαφυγή αερίου για την προστασία της επιφάνειας και ιδίως ε, τα ε, υπόγεια ύδατα. Ουσιαστικά το σημαντικό είναι να προσέξει κανείς το σχεδιασμό του φρέατος, το σχεδιασμό της γεώτρησης. Υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές, ε, από τις πιο αυστηρές είναι οι ευρωπαϊκές. Τηρούμε όλες αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Έχουμε τρία περιβλήματα, τρία casing, ένα εξωτερικό, ένα ενδιάμεσο που στη Βόρεια Αμερική Συνήθω δεν χρησιμοποιείται και έχουμε και το τρίτο περίλημα, το τρίτο κέλυφος ε, που προστατεύει πάρα πολύ ε, καλά. Πριν έχουμε το σχηματισμό των τρόγων ανθράκων. Υπάρχουν λοιπόν αυτά τα περιβαλλοντικά ζητήματα, υπάρχει ζήτημα εμπιστοσύνη, όπω είπα, τη κοινή γνώμη. Πολλοί δεν καταλαβαίνουν τι κάνουμε, είναι κάτι καινούριο για πολλοί κόσμο και γι' αυτό πρέπει να έχουμε πλήρη δημοσιοποίηση των στοιχείων. Εμείς ε, δημοσιοποιούμε στην ιστοσελίδα μας ε, όλα τα υγρά τα οποία χρησιμοποιούνται, τις χημικές ουσίες, ε, Όλα, όλα αναφέρονται, είτε τα χημικά που χρησιμοποιούμε είτε για την γεώτρηση είτε για την αρωμάτωση. Και γενικά είμαστε υπέρ της ανοιχτής, της διαφάνειας με όλους. Και έχουμε ε, πολλούς επισκέπτες, ε, μέχρι και κατοίκου της περιοχής, αγρότες και φυσικά και εξωματικούς τη κυβέρνηση που έχουν ε, επισκεφθεί, χιλιάδες τέτοιε επισκέψεις έχουν γίνει στις εγκαταστάσει μας, όπου τους δείχνουμε ακριβώ τι κάνουμε και ποιε ασφαλιστικές δικλείδες έχουμε για να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Για τη χρήση του νερού μίλησαν πολύ, πόσο δηλαδή νερό χρησιμοποιείται για την παραγωγή ισχυστολιθικού φυσικού αερίου. Αν δείτε τι γίνεται, πόσο αέριο χρησιμοποιούμε για την παραγωγή ισχύω είναι πολύ λιγότερο σε σχέση με αυτό που χρησιμοποιείται από έναν ε, πυρηνικό σταθμό ή από ένα εργοστάσιο άνθρακα. Σίγουρα λοιπόν καταναλώνουμε λιγότερο νερό σε σχέση με άλλα ενεργειακά ε, συστήματα. Πολλοί φαίνεται όμως να νομίζουν ότι όταν κάποιος κάνει αυτή την ε, ρογμάτωση έχει συνεχείς ροές ε, νερού. Αλλά όχι, μία φορά γίνεται η ρογμάτωση. Δεν γίνεται για μακρά χρονική περίοδο, αλλά ε, το νερό χρησιμοποιείται για ένα πολύ μικρή χρονική περίοδο. Και ανακύκλωση του νερού είναι κάτι το οποίο γίνεται κατά κανόνα. Είναι πολύ πιο οικονομικό να το ανακυκλώσουμε το νερό στο δυνατό σε μεγαλύτερη ποσότητα και έτσι είναι πολύ πιο οικονομικό προσπαθούμε έστω και κοντά στο 100% αν δεν μπορούμε 100% να το ανακυκλώσουμε. Νομίζω ότι αυτό κάνουν και περισσότερες σύγχρονες εταιρείε. Έχουμε τα green flowbacks, πράσινη επιστροφή ροής, μετά δηλαδή την ε, υδρορογμάτωση. Ούτε έχουμε εξαέρωση του αερίου στο στην ατμόσφαιρα, το μεταφέρουμε στη σχετική εγκατάσταση καύσης το συντομότερο δυνατό και γίνεται πολύ καλύτερο διαχωρισμός ε, του αερίου και προσπαθούμε να λεξιτοποιήσουμε ε, την έκκληση ε, αερίου στην ατμόσφαιρα. Δεν θέλουμε να εκλειθεί αέριο στην ατμόσφαιρα, δεν θέλουμε να έχουμε διαφυγές, δεν θέλουμε να έχουμε εξαέρωση. Όσο το δυνατόν λιγότερο είναι το αέριο το οποίο δεν περνάει στην όλη αυτή αλυσίδα παραγωγής του αερίου. Εδώ βλέπετε τα χημικά που χρησιμοποιούμε και τις ποσότητες. Είτε κάνουμε ρογμάτωση και βλέπετε και τις διάφορες επιγές, βλέπετε τα κελίφη και εδώ βλέπετε και ένα ground gas monitor, ένα μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιούμε εδώ βλέπετε τον ε, διαχωριστή, το separator, δεν ξέρω αν έχετε δει ποτέ, και αυτές τις δεξαμενές ε, flow back. Και βλέπετε και τη μεμβράνη αυτή, την διαπερατή που οτιδήποτε δηλαδή ε, περάσει προς το έδαφος συγκρατείται στη μεμβράνη αυτή. και μετά μπορούμε να διαθέσουμε με το σωστό τρόπο αυτή τη μεμβράνη. Κάτι άλλο το οποίο συμβαίνει συχνά είναι ότι δεν έχουμε επαρκή σπόρους. Για το σχιστολιφικό σκάρο δεν θα έπρεπε να ανησυχούμε ουσιαστικά. Μόλι ολοκληρώσαμε ε, κάποιε αδρέ εκτιμήσει, μόνο και μόνο για τη λεκάνη του Μπόλαντ ε, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, με 200 TCF. Αυτό ε, σημαίνει ότι υπάρχει αυτό το αέριο, όχι ότι θα το ανακτήσουμε όλο αυτό, όλη αυτή την ποσότητα. Θα είναι πολύ χαμηλότερη η ποσότητα που θα ανακτηθεί, αυτό θα το γνωρίζουμε όταν θα έχουμε περισσότερες γεωτρήσεις, θα έχουμε κάνει περισσότερες υδρορογματώσεις και θα μπορούμε να κάνουμε και τους σχετικούς ελέγχους για να δούμε πόσο αέριο μπορεί να παραχθεί. Ε, υπάρχουν πάντως πολλές ε, αναλύσεις, ε, core και cutting ε, και σεισμικές μελέτες κάνουμε σε δύο διαστάσεις, οπότε ουσιαστικά μπορούμε να είμαστε αρκετά αισιόδοξοι. 200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι που έχουμε, ε, μάλλον 1.200 ε, ε, τετραγωνικά χιλιόμετρα είναι που έχουμε και βλέπετε και το σχετικό διάγραμμα. Υπάρχει και μία μελέτη που έχει γίνει για τον οικονομικό αντίκτυπο 400 φρεάτια είδαμε, 400 φρεάτια 400 ε, ουσιαστικά χώροι με 10 φρεάτια ο καθένας. Ε, για 9 χρόνια θα είχαμε 10 ε, γεωτρήσεις που θα έπρεπε να γίνουν και θα υπήρχαν και πολλές θέσεις εργασίας. 5.600 συγκεκριμένα ε, πλήρους απασχόληση, δύναμος πλήρους απασχόλησης. Και θα είχαμε και την εχμή από το 2016 στο 2019. Έτσι θα μπορούσαμε να είχαμε έσοδα φορολογικά γύρω στα 6 με 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα της ανεξάρτητης μελέτης της Regeneris Consulting. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να ε, είμαστε οικονομικά αποδοτικοί. Τώρα γνωρίζουμε πού υπάρχει το αέριο αυτό, ξέρουμε που μπορούμε να κάνουμε τις γεωτρήσεις και τις εξορίξεις με ασφάλεια, αποτελεσματικά, που μπορούμε να κάνουμε την υδραυλική ρογμάτωση. Βλέπετε το φλερ, βλέπετε αυτή την εγκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι κλειστό, δηλαδή ουσιαστικά δεν βλέπετε τη φλόγα δηλαδή, αλλά βλέπετε, ε, εκεί γίνεται η διαδικασία της καύσης και θα αξιολογήσουμε και θα δούμε πόσο φυσικό αέριο μπορεί να παραχθεί σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τους ομιλητές και θα αλλάξουμε λίγο για να έρθουν οι επόμενοι τρεις ομιλητές. Ευχαριστώ.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 Okay. Darf noch mal bitten, Παρακαλώ και πάλι προσπαθήστε όλοι να τηρήσετε τον προκαθορισμένο χρόνο γιατί ο χρόνος τρέχει και δεν θα μας μείνει ώρα για ερωτήσεις. Δεν ε, είμαι κακός που τα λέω αυτά. Τα είπαμε και από πριν, τα συμφωνήσαμε και παρακαλώ να τηρηθούν οι χρόνοι. Προχωρούμε τώρα στις μελλοντικές τεχνολογικές εξελίξεις, ε, δυνατότητες. Έχουμε τρεις ομιλητές που κατέχουν βεβαίως διαφορετικές θέσεις. Ο πρώτος ομιλητής μας είναι ο κύριος Ρόμπερτ Χάουαρθ, καθηγητής από τη Νέα Υόρκη. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας μιλήσω. Χαίρομαι πολύ που ήρθα από τις Ηνωμένε Πολιτείε, Θα ήθελα να αναφερθώ σε διάφορα θέματα ως επιστήμον, να δούμε δηλαδή τι βλέπουμε τώρα να γίνεται στη ΣΥΠΑ. Θα κάνουμε και ανασκόπηση περιβαλλοντικών θεμάτων και θα επικεντρώσουμε στην δική μας δουλειά εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με το σχιστολιθικό αέριο. Προσπερνώ μερικά εδώ θα ήθελα να διαφωνήσω λίγο με την τελευταία ομιλία, αλλά θεωρώ ότι οι περισσότεροι από εμά που παρακολουθούν τις εξελίξεις της ΕΠΑ, η ανάπτυξη του συστολιθικού αερίου είναι καινούρια τεχνολογία η οποία απαιτεί υψηλής εξειδίκευσης, οριζόντια, γεώτρηση ε, μεγάλων αποστάσεων και μεγάλες ποσότητες νερού για την υδρορογμάτωση. Η τελευταία χρησιμοποιείται εδώ και καιρό και στη, στον κλάδο αερίου και πετρελαίου και στη ΣΥΠΑ που και στη, στα συμβατικά ε, φρεάτια έκαναν ε, ρογμάτωση αλλά όχι με τον τρόπο που απαιτεί το συστολιθικό γιατί τώρα ε, κατά μέσον όρο χρησιμοποιούνται 20 εκατομμύρια νερό για ένα φρεάτιο 12 με 16 ε, πηγάδια υπάρχουν ανά πάντ, πολύ νερό, σε σχέση με τις συμβατικές ρογματώσεις που χρησιμοποιούσαν κατά μέσον όρο, όχι, κατά μέγιστον 300.000 λίτρα. Οπότε είναι πολύ εντατική διαδικασία, πολύ νερό ξαναγυρίζει στην επιφάνεια και υλικά πηγαίνουν προς τα κάτω και άλλα αφαιρούνται με τις επιφανειοδραστικές ουσίες από το νερό. Επειδή είναι καινούργια διαδικασία, στο Τέξας αναπτύχθηκε πριν από 15 χρόνια, ε, όπως ακούσατε, έχουν στο Burnett Shell, ε, για τους, εκεί έχει αναπτυχθεί. Για τους άλλους είναι νέα τεχνολογία, ε, των τριών, τεσσάρων, maximum πέντε ετών. Ε, είναι καινούργια και στους εκτός ΙΠΑ και στις ΙΠΑ. Είναι καινούρια μέθοδος και για την επιστημονική κοινότητα. Δηλαδή ακόμα δεν έχει γίνει πλήρης περιβαλλοντική ανάλυση. Εξελίσσεται τώρα. Οι πρώτες, ε, τα πρώτα άρθρα στην επιστημονική ε, βιβλιογραφία τους 6-7 τελευταίους μήνες δημοσιεύτηκαν. Θα πάω πολύ γρήγορα ε, τώρα. Η τοπική ατμοσφαιρική ρήπανση είναι μεγάλο πρόβλημα για το όζον από τα μηχανήματα, το βενζόλιο, υδρογονάνθρακες, ε, αλογονωμένη. Αυτά είναι γνωστά όμως. Η ρήπανση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων λαμβάνει χώρα και το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εντοπίσει μέχρι τώρα είναι τι γίνεται με τα απόβλητα που ε, έρχονται στην επιφάνεια από την ρογμάτωση. Γίνεται ανακύκλωση, αλλά ε, όχι σε όλα υπάρχουν κάποιες ε, λάθος αναφορές από την περασμένη άνοιξη, από την Πενσιλβανία, που έλεγαν ότι όλα τα ανακυκλώνουν. Ο, έγινε σωστός υπολογισμός και μόνο το 2,6% ε, ανακυκλώνεται 30% δεν ξέρουμε που πάει, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε και τα υπόλοιπα από το 2010 στην Πενσιλβανία πήγαινε σε δημοτικές εγκαταστάσεις ε, ε, βιολογικού καθαρισμού. Δημιουργήθηκαν προβλήματα. Τώρα απαγορεύτηκε αυτό στην Πενσιλβανία. Αυτό που κάνει η βιομηχανία τώρα δεν είναι σαφές, αλλά δεν ε, είδα μεγάλη αύξηση της ανακύκλωσης. Η ανακύκλωση είναι πολύ μικρής κλίμακας. Κάτι άλλο τώρα, ε, μεθάνιο, αέριο του θερμοκηπίου, ρήπανση των ε, υπογείων υδάτων. Δεν ξέρω αν έχετε δει την ταινία Gasland που λένε ότι είναι... Ε, πολύ ε, λίγο σκανδαλοθυρική, τη λένε μερικοί. Ε, τώρα, τι γίνεται με το μεθάνιο, είναι δύσκολο να ξέρουμε εδώ ας πούμε τι ακριβώς γίνεται. Λένε ότι δημιουργούνται προβλήματα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία και αυτή είναι μια εργασία που δημοσιεύτηκε ε, στα πρακτικά της ε, Ακαδημίας Επιστημών τον περασμένο Μάιο. Ε, έκαναν δειγματοληψία στο μεθάνιο, το οποίο είναι στη, στα πηγάδια ποσίμου νερού κοντά στο φρεάτιο του αερίου. Αν είμαστε σε απόσταση ενός χιλιόμετρου μπορεί να υπάρχει μεθάνιο, αλλά όχι πολύ και φαίνεται ότι είναι φυσικό ε, μεθάνιο, όχι από τη βιομηχανία. Αν όμως είμαστε ε, ένα χιλιόμετρο μακριά και αυτό συμβαίνει και στο Μαρσέλο Σέιλ και στη Νέα Υόρκη και στην Πενσιλβανία ε, μπορεί κατά 75% να έχουμε υψηλά επίπεδα μεθανίου και στο Μαρσέλ Σέιλ έχουμε έντονη βιομηχανική ε, δραστηριότητα. Έτσι λοιπόν ε, μπορεί να ακούσει η ταινία το, το φιλμ σκανδαλοθυρικό, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τη βιομηχανία. Αυτά τα προσπερνώ, είναι της βιομηχανίας διαφάνεια που δείχνει ότι αν δεν γίνει καλή δουλειά στη γεώτρηση ε, υπάρχει μηχανισμός να, που διοχετεύει το μεθάνιο στον υδροφόρο ορίζοντα ε, Επίση, μια μελέτη δείχνει ότι ρήπανση υπάρχει και σε μεγάλη κλίμακα. Για να δούμε τώρα τα, τα, τις αερίων του θερμοκηπίου. Αυτή είναι η δική μας έρευνα. Ε, είναι ένα ερευνητικό θέμα που το αρχίσαμε πριν από δύο χρόνια με συναδέλφους και θέλαμε να κάνουμε πλήρη ανάλυση του κύκλου ζωής του και του αποτυπώματος του σχιστολιθικού αερίου. Ε, αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη ε, μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Peer Review Journal τον Απρίλιο και αυτή είναι μια περίληψη. Αυτό έχει ανατυπωθεί από το, ένα άρθρο στο Nature πριν από τρεις εβδομάδες, αν σας ενδιαφέρει, ε, σχόλια για τα γενικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Ε, εδώ βλέπουμε το διοξίδιο του άνθρακα, αριστερά το συστολιθικό με περιορισμένη διήστηση, το συμβατικό ε, και το δίζελ κάψιμο. Ε, βλέπουμε επίσης ανάμορφη ενέργεια σε πόσο διοξίδιο του άνθρακα παράγεται. Το φυσικό αέριο και το συστολιθικό εκλείουν λιγότερο ε, διοξίδιο του άνθρακα. Είναι καθαρά υπό αυτή την έννοια. Είδαμε όμω και το μεθάνιο. Το φυσικό αέριο αποτελείται από μεθάνιο επιτοπλίστων που είναι πολύ ισχυρό αέριο θερμοκηπίου και υπάρχουν μικρές ε, διαρροέ ε, και οι μικρές διαρροές στην ατμόσφαιρα συμβάλλουν πολύ στην αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου. Και αυτή η μελέτη δείχνει εδώ με το ροζ κόκκινο χρώμα την επιρροή του μεθανίου στο αποτύπωμα των ε, αερίων θερμοκηπίου ε, σε σχέση με την ισοδυναμία ε, του διοξιδίου του άνθρακα. Και βλέπουμε εδώ και το στοιχεία σχετικά με το χρόνο μετά την έκκληση. Εδώ με βάση τα δικά μας στοιχεία και εκτιμήσεις βλέπουμε ότι και όταν είναι χαμηλές περιορισμένες οι εκτιμήσεις για τις εκπομπές συστολιθικού μεθανίου με τις καλύτερες διαθέσιμες τεχνολογίες που δεν είναι απαραίτητα αυτές που χρησιμοποιούν στη βιομηχανία ακόμα και από αυτές τις συνθήκες είναι μεγαλύτερο το αποτύπωμα στο αέριο θερμοκηπίου από ότι στον άνθρακα ε, ή τα συμβατικά αέρια. Ε, τα υψηλότερα, αν κάνουμε εκτιμήσεις προς τα πάνω, ε, χειροτερεύουν τα πράγματα. Η, με βάση τις πληροφορίες που οι πληροφορίες μας είναι περιορισμένες ακόμα για τέτοιες μελέτες, η τεχμηρίωση δεν είναι μεγάλη, αλλά βάζουμε κάτω τις ε, καλύτερες πληροφορίες που μπορούμε να συγκεντρώσουμε για τη μελέτη αυτή. Θα μπω σε λεπτομέρειε αν με ρωτήσετε. Τώρα, σχετικά με το χρονικό ορίζοντα. Εδώ στο πάνω, στην πάνω διαφάνεια είναι αυτά που σας έδειξα, ε, τα διάφορα ε, έτη και από το περιοδικό Nature. Εδώ ο χρονικός ορίζοντας 20 ετή... σε σχέση με το αποτύπωμα των αερίων θερμοκηπίου. Κάτω είναι χρονικό ορίζον 100 χρόνια ε, ολοκληρωμένο. Εδώ μειώνεται η επίδραση του μεθανίου. Γιατί? Γιατί σε σχέση με το διοξίδιο του άνθρακα δεν μένει το μεθάνιο τόσο πολύ. Έχει πολυματικό χρόνο παραμονή, περίπου 10 χρόνια. Ενώ είναι 100 χρόνια ο αντίστοιχο χρόνο παραμονή για το διοξίδιο. Έτσι λοιπόν βράχει πρόθεσμα είναι μεγάλο το πρόβλημα για το, ε, από το μεθάνιο, το οποίο αργότερα ε, μειώνεται. Ε, οπότε στα 100 χρόνια είναι περίπου το ίδιο όπως το αποτύπωμα του διοξίδιου του άνθρακα. Θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντική η μικρότερη χρονική κλίμακα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί οι επιστήμονες, ειδικοί για το κλίμα, ε, ανησυχούν πάρα πολύ ότι είμαστε σε οριακό σημείο ως ε, πλανήτης Γη τις επόμενες δεκαετίες τα 30, 40, 50 χρόνια, όχι 100 και 150. Ένα οριακό σημείο που μπορεί να μας γυρίσει σε εναλλακτικό κλιματικό σύστημα, πάρα πολύ δυσμενές από την άποψη της αηφορίας, της γεωργίας και άλλα θέματα της κοινωνίας. Και όταν πάμε σε αυτό το εναλλακτικό σύστημα του κλίματος, δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στο σημείο εκκινήσεώς μας. Θέλουμε να αποφύγουμε λοιπόν ε, οποιαδήποτε υπερθέρμανση που θα μας οδηγήσει σε κάτι τέτοιο γιατί αλλάζουν οι, ε, αλλάζει η κατάσταση των υδάτων στους ωκεανούς, η κυκλοφορία των υδάτων, ε, γιατί είναι πάρα πολύ ενσυχητικό το πώς προσλαμβάνει το διοξίδιο του άνθρακα ή η θέρμανση των ακτικών περιοχών, οπότε και εκεί θα υπάρχει έκκληση μεθανίου ε, σε μεγάλη επιτάχυνση και αν συμβεί αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντιστραφεί. Πρέπει να προσέχουμε λοιπόν πολύ όχι μόνο τις μακροπρόθεσμες ε, ε, εξελίξεις αλλά και τις βραχυπρόθεσμες σε ό,τι αφορά το αποτύπωμα και εκεί το συστολιθικό είναι πάρα πολύ ε, δυσμενές αρνητικό κάψιμο. Τον Απρίλιο είχαμε μια την πρώτη περιεκτική μελέτη, peer-reviewed, ε, που έχει εξεταστεί από ομολόγους και αξιολογηθεί. Από τότε που εξεδόθη η μελέτη ακολούθησαν κι άλλες. Ακούσαμε στοιχεία από προηγούμενε ομιλίε. Η νέα μελέτη από, τον οργανισμό, από την Υπηρεσία Ατομική Ενέργεια δεν την έχω δει. Γνωρίζω άλλε όμω που έχουν ε, κυκλοφορήσει μετά από τη δική μα. Ε, μία είναι του David Hughes, θέλω να αναφέρω, προ... από τον Καναδά, γεωλόγο ε, υπάρχουν άλλοι που παίρνουν παρόμοια ε, θέση. Ε, έχουμε και έναν παρόντα μοιάζει με, την, ε, με μια άλλη παγκόσμια μελέτη. Υπάρχει και μια μελέτη από το Weekly. Ε, τον Αύγουστο είχαμε δύο μελέτες ε, που, που κυκλοφόρησαν για να δούμε πώς, τι αποτελέσματα δίνουν. Εδώ θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά θέλω να ξέρετε ότι εμείς εξετάζουμε τις λεπτομέρειες, γιατί η λεπτομέρεια μετράει. Να σας πω λοιπόν τις διαφορές στις μελέτες η πρώτη στήλη εδώ είναι η δικά μας μελέτη σε σχέση με άλλες. Ε, βλέπετε εδώ τη χρονική κλίμακα. Βλέπουμε και τη μικρότερη χρονική κλίμακα και τη μακρότερη ε, και η εργασία Wigley και η εργασία Hughes επίσης. Οι άλλες εξέτασαν ε, μόνο τα 100 χρόνια, πράγμα που υποτιμά τη σημασία του μεθανίου. Μετά έχουμε το θέρμανση παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας και βλέπουμε πώς συγκρίνονται τα ε, διάφορα στοιχεία. 33-105 ε, βραχύτερη και μακρότερη χρονική κλίμακα. Αυτά είναι τα τελευταία επιστημονικά μοντέλα που δημοσιεύτηκαν στο Science, το περιοδικό αυτό, το Νοέμβριο του 2009. Ο Wigley δεν χρησιμοποιεί τέτοια μοντέλα, έχει ένα πιο εκλεπτισμένο ατμοσφαιρικό μοντέλο ε, οι άλλες μελέτες, ο Χιούς ακολουθεί την ίδια μελέτη, οι άλλοι χρησιμοποιούν το 25 που είναι η ανάλυση των 100 ετών που πάλι υποτιμά το μεθάνιο, αναφέρεται ε, και τελευταία σε μια ανάλυση της ICC. Το, η νέα εκτίμηση IPC δίνει μεγαλύτερα, θα δώσει μεγαλύτερα νούμερα όταν εκδοθεί. Ε, επίσης, ε, θερμότητα και ηλεκτρική ενέργεια. Ω ε, επιτοπλίστων για την παραγωγή θερμότητα χρησιμοποιείται στη ΣΥΠΟ Ο Χιούζ εξετάζει και τα δύο. Όλοι οι άλλοι κοίταξαν μόνο την παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια. Ε, και εμεί κοιτάξαμε τα δύο βέβαια. Μετά είδαμε διάφορες εκτιμήσεις για τις εκπομπές μεθανίου. Έχουμε εδώ διαφοροποίηση σε σχέση ε, με τις ε, τιμές που χρησιμοποιούμε. Διάφορες μελέτες χρησιμοποιούν ε, νούμερα δύο-τρεις φορές χαμηλότερα από αυτά που λέει η IPA και σε σύγκριση με την διαφυγή μεθανίου από τον άνθρακα πάλι τα στοιχεία μας είναι κοντά σε αυτά που δίνει η EPA. Άλλοι στηρίζονται σε πεπαλαιωμένα στοιχεία από τη βιβλιογραφία. Τα μπλε στοιχεία εδώ δείχνουν ότι είναι χειρό, χειρότερο από τον άνθρακα ε, το σχιστολιθικό σε, 15, σε χρονικό ορίζοντα 15 ετών, είτε για ε, ηλεκτρική ενέργεια ή θερμότητα. Ε, το κόκκινο εξετάζει τα 100 χρόνια και λέει ότι ναι, είναι καλύτερο το σχιστολιθικό αέριο από τον άνθρακα. για λόγους χρόνου θα σας δείξω εδώ κάτι. Ακούσατε τις εκτιμήσεις το συστολιθικό και τι ξέρουμε και τι δεν ξέρουμε. Η εισαγωγή από την IEA ήταν πάρα πολύ ε, καλή. Εγώ θα ήθελα να πω ότι στις είπα οι εκτιμήσεις μας ε, μειώθηκαν πάρα πολύ τα, τις τελευταίες 5-6 εβδομάδες μετά από μια άλλη έρευνα γεωλογική του Μαρσέλου Σέλιο, που είναι το μεγαλύτερο κοίτασμα, που δείχνει ότι οι προηγούμενε εκτιμήσει από το Υπουργείο Επιστήμης ήταν πέντε φορέ υψηλότερα. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ε, στοιχεία τα οποία ενδεχομένω να ήταν ε, γνωστά και παλιότερα. Ε, πάμε στα συμπεράσματα. Είναι καινούριο, είναι πειραματικό το συστηματικό αέριο. Ε, υπάρχουν πολλοί περιβαλλοντικοί κίνδυνοι που δεν έχουν ακόμη ε, αντιμετωπιστεί ή γίνει πλήρως κατανοητή. Το αποτύπωμα των αερίων θερμοκηπίου είναι μεγαλύτερο από άλλα ορυκτά καύσιμα αν δούμε 50 χρόνια ή λιγότερα ως χρονική κλίμακα και οι πόροι μπορεί να είναι λιγότεροι από ό,τι ισχυρίζονται οι υπέρμαχοι αυτή τη μορφή ενέργεια. Οπότε εδώ πραγματικά θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ προσεκτικά. Ευχαριστώ για την προσοχή σα και για την ευκαιρία που μου δώσατε να έρθω σήμερα. Και τώρα ο κύριος Πίστρε, καθηγητής υδρογεωλογίας από το Πανεπιστήμιο του Μομπελιέ. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Εγώ είμαι καθηγητής της υδρογεωλογίας στο Μοντελιέ, στο και θα επικεντρώσω την ε, τοποθέτησή μου στην ε, διατήρηση των φυσικών μας πόρων μέσα από αυτού του είδους τα εγχειρήματα. Εμείς έχουμε τρεις προκλήσεις. Για την σχιστολιθική γεώτρηση έχουμε την ποιότητα, όπου έχουμε δύο προβλήματα, το θέμα της άμεσης ρήπανσης και της έμεσης ρήπανσης. Και θα σας το εξηγήσω. Για τους, απαραίτη, για τους απαραίτητους ε, όγκους, 10 με 20 χιλιάδες τόνους, Εμείς ε, λοιπόν ε, όταν περνάμε από την επιφάνεια ψάχνουμε τα υπόγεια ύδατα. Τα επιφανειακά ύδατα αρκούν, αλλά όταν μεταφέρουμε αυτά τα ύδατα στο χώρο της γεώτρησης είτε με φορτηγό είτε με σωλήνες, να ας πούμε δείτε 1800 κυβικά το δευτερόλεπτο είναι ο ροδανός άμα δούμε το πόσο χρησιμοποιούμε εμείς στο, στην γεώτρηση, αυτό δεν είναι τίποτα με τις μεγάλες ροές των ποταμών. Έχουμε λοιπόν δύο δυνατότητες. Είτε να έχουμε Είτε λοιπόν να έχουμε μία παράλληλη γεώτρηση και να χρησιμοποιήσουμε είδωρ το οποίο χρησιμοποιείται για, άλλες, ε, για άλλα πράγματα, ας πούμε ποτιστικά ύδατα να τα χρησιμοποιήσουμε ή φρεάτια να χρησιμοποιήσουμε ε, νερό από φρεάτια τα οποία δεν έχουμε ακόμη εκμεταλλευτεί. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε υδραυλικές συνδέσεις μεταξύ των δύο και να έχουμε προβλήματα σε αυτό το επίπεδο. Το συμπέρασμά μου είναι ότι μπορούμε να έχουμε λύσεις ε, για την ε, διαχείριση των διαφόρων ποσοτήτων χωρίς πλάβες ε, για το περιβάλλον. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Να δούμε τώρα την άμεση ρήπανση του ύδατος. Εμείς έχουμε μία επιφανειακή ρήπανση που αφορά στα επιφανειακά ύδατα, αλλά μετά έχουμε και την απορρόφηση η οποία μπορεί να επηρεάσει τα υπόγεια ύδατα. Μπορούμε να έχουμε επίσης από ατύχημα τη, τη ρήπανση φρεατίων συλλογής ύδατος. Πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν τέτοιου είδους εκχυλήσεις. Και μετά έχουμε και τη ρήπανση που μπορεί να προκληθεί από τη διαφυγή βιομηχανικών ουσιών, βιομηχανικών υγρών ε, γύρω από την πλατφόρμα. Επίσης μπορούμε να έχουμε διασωλήνωση της γεώτρησης η οποία να είναι ελαττωματική. Μπορείτε να δείτε εδώ στη διαφάνεια τι προβλήματα μπορούν να προκύψουν. Προϊόντα τα οποία μπορούν να διαφύγουν μέσω από, την, ε, από το σύστημα γεώτρησης ε, και να ρηπάνουν τα υπόγεια ύδατα. Μετά έχουμε τον κακό έλεγχο. Έχουμε ας πούμε τις σχισμές από την υδρο... υδραυλική γεώτρηση που μπορούν να επηρεάσουν τα διάφορα στρώματα. Άλλα, προβλήματα τα οποία συνδέονται εν δυνάμει με όλα αυτά είναι το να ανοίξουμε ακόμη παραπάνω τις σχισμές στα στρώματα σχιστολίθου και να επιτρέψουμε ουσίες να διαφύγουν προς την επιφάνεια. Μετά έχουμε τα εγκαταλ... τις εγκαταλελειμμένες γεωτρήσεις, τα εγκαταλελειμμένα φρεάτια, όπου μπορούμε να έχουμε διασύνδεση μεταξύ των ε, διαφόρων ε, φρεατίων υπογείων υδάτων με αυτά τα φρεάτια και να έχουμε διαφυγές. Υπάρχουν λύσεις για να μειώσουμε τους κινδύνους, αλλά είναι δυσεφάρμοστες. Ανάλογα βέβαια με τις γεωλογικές συνθήκες. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο δεν αναφέρεται συχνά, έχουμε μία δημοσίευση που αφορά στο πρόβλημα, είναι η έμεση ρήπανση. Αυτό μπορεί να αφορά και στην επιφάνεια αλλά και να προέρχεται μάλλον από την επιφάνεια αλλά και από το βάθος, από το βυθό. Εμείς μπορεί να έχουμε πλούσιες ε, οργανικές ουσίες ε, και, αργυ, άργυλο που μπορεί να εγκλείει ραδιενεργές ουσίες, μέταλλα ή μεταλλοειδείς ουσίες, με, μετάλλιουμ κλπ. Ουράνιο, μόλιβδο, ράδιουμ. Για παράδειγμα, στη Νότιο Γαλλία έχουμε Έχουμε μία φλέβα σχιστόλιθου η οποία βρισκόταν σε παλιά μεταλλεία ουρανίου. Δηλαδή μπορεί κάλλιστα να περικλεί, να περικλεί στη διαστρωμάτωσή του ουράνιο. Τώρα λόγω της χημικής ισορροπίας και σύνθεσης αυτών των ουσιών μένουν, έχουν, βρίσκονται σε ακινησία. Όταν εμείς πηγαίνουμε να κάνουμε την εξόριξη και αρχίσουμε να αντλούμε όλα αυτά τα στοιχεία, απολευθερώνονται και μπορούν να βγουν στην επιφάνεια. Επίσης, έχουμε και τις, έχουμε και τα αέρια τα οποία μπορούν να διαφύγουν και να ρυπάνουν επιφανειακά τα διάφορα στρώματα. Η υδραυλική εξόριξη θέλει να επιτρέψει πιο εύκολα την διαφυγή του αερίου. Αλλά όμως έχουμε εμείς αυτές τις μεταλλικές ή ραδι... ραδιενεργές ουσίες που μπορούν να διαφύγουν από αυτά τα στρώματα και αν αλλάξουν και άμα έχουμε δυσμενείς γεωλογικές συνθήκες μπορούν όλες αυτές οι ουσίες μπορούν να φύγουν στην επιφάνεια κυρίως όταν έχουμε βαθιές ρογμές. Ας πούμε αν πάρετε ένα μικρό μπουκάλι νερό, θα έχετε μπροστά σας, θα δείτε ότι αυτό το νερό το έχουν, ε, το έχουν πάρει από μία πηγή που βρίσκεται σε 1600 μέτρα βάθους κάτω από τη γη. Και αυτό αποτελεί εγγύηση της καθαρότητας του ύδατος. υπάρχουν ρίσκα γεωλογικού χαρακτήρα και δεν υπάρχουν τεχνικές λύσεις. Ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε επεξεργασία των υγρών αποβλήτων Δεν μπορώ να φανταστώ εγώ καμιά άλλη λύση. Έχετε εδώ τώρα το χάρτη της Γαλλίας με τις τρεις ε, μεγάλες λεκάνες όπου θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε το σχιστολιθικό ε, ε, φυσικό αέριο. Έχετε εδώ την νότιο-ανατολική λεκάνη, μεσογειακό κλίμα και με λίγο νερό το καλοκαίρι. Και έχουμε καρστικές ε, πηγές ε, ε, υδάτων. Επίσης πρόκειται για ταλαιπωρημένη γεωλογικά περιοχή διότι έχουμε βαθιές ρογμές και έχουμε αυτές τις ρογμές οι οποίες είναι γεμάτες είτε με νερό είτε με διοξείδιο του άνθρακα. Βλέπετε τώρα εδώ με πράσινο και με κίτρινο τα διάφορα υπόγεια ύδατα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, έχουν στρατηγική σημασία για τον πληθυσμό. Έχουμε εδώ πόσιμα ύδατα Και βλέπετε ότι υπάρχει πολλές φορές εδώ πάνω στο χάρτη επικάλυψη μεταξύ των αντιών εκμετάλλευσης σχιστόλιθου με τις πηγές νερού. Έχετε με μπλε επίσης τις πηγές νερού, πόσιμου νερού, που επικαλύπτουν τους τόπους εκμετάλλευσης του σχιστόλιθου. Το νερό αυτό το παίρνουμε μέσα από ρήγματα 2.000 μέτρων και άμα το δείτε δηλαδή από κοντά βλέπετε τη ρογμή η οποία φτάνει μέχρι την πηγή βλέπετε το νερό ότι με τα κόκκινα βέλη ότι ανεβαίνει μέσα από αυτήν τη ρογμή και βγαίνει στην επιφάνεια. Αν αλλάξουμε εμείς τις παραμέτρους αυτών των φρεατίων, ραδιοϊσόπατα, ε, ισο, <laughs> ραδιοϊσότοπα και οι μεταλλούχες ουσίες απολευθερώνονται, βγαίνουν στην επιφάνεια. Τώρα εγώ δεν ξέρω αν η τεχνολογική πρόοδος θα μας επιτρέψει να μειώσουμε αυτόν τον κίνδυνο της ρήπασης του πόσιμου ύδατος. Τώρα, για την κάθε τοποθεσία εκμετάλλευσης χρειάζεται μία απαραίτητη υδρογεωλογική μελέτη για να αξιολογηθεί ο κίνδυνος και να μπορέσουμε να εξισορροπήσουμε το κέρδος ωφέλεια θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό για το τι θα συμβεί στο οικοσύστημα κατά την εκμετάλλευση αλλά και μετά την εκμετάλλευση διότι όπως σας εξήγησα η δυναμική των υπογείων υδάτων ε, είναι μια τεράστια διαδικασία, μακρόχρονη διαδικασία. Εμείς κάλλιστα μπορούμε να κλείσουμε μια πλατφόρμα εκμετάλλευσης, τότε το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ράινικε από το Ινστιτούτο ε, Μηχανολογικού Σχεδιασμού Πετρελαίου από το Κλάουσταλ. Ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω εδώ σε εσάς Λέγομαι Κουρτ Ράινικε, είμαι από το, το Πολυτεχνείο του Κλάουσταλ. Εδώ και χρόνια δουλεύω στην πετρελαιοβιομηχανία. Τη δεκαετία του 70 και 80 ασχολούμαι με ρογμάτωση και τα τελευταία χρόνια είμαι στο Κλάουσταλ στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ε, θα μιλήσω για το συστολιθικό αέριο, εγώ θα πω για την ανάπτυξή του και για περιβαλλοντικά θέματα. Ε, το σχιστολιθικό αέριο είναι μη συμβατικό, συμπαγές αέριο, αλλά δεν είναι το αέριο μη συμβατικό, η τεχνολογία είναι μη συμβατική για την παραγωγή του. δηλαδή πολλές φορές η ροή δημιουργεί προβλήματα και γι' αυτό χρειάζονται μη συμβατικές τεχνολογίες. Θα σας δείξω το δυναμικό και την ε, ε, ε, ικανότητα ροής, το βαθμό ροής. Εδώ βλέπουμε μια σημαντική δεξαμενή. Βλέπετε ότι εκεί είναι καλές ιδιότητες ροής, ρεολογικές ιδιότητες σε σχέση με άλλες. Οι ιδιότητες ενός πεζοδρομίου σκυροδέματος ενδιαφέρουν επίσης σε ό,τι αφορά την ε, διαπερατότητα. Οι δεξαμενές ε, μη συμβατικού αερίου επίσης είναι διαφορετικές από των συμβατικών. Είναι πολύ χαμηλή η διαπερατότητα εκεί. Χρειάζονται λοιπόν άλλες τεχνικές. Αλλά οι δυνατότητες που μας δίνουν είναι τεράστιες. Το σχιστολιθικό είναι στη Βόρεια Γερμανία, στη Λεκάνη εκεί, στο Φίλτεν, Ποσειδονία. Βλέπουμε εδώ ε, αυτές τις, ε, αυτά τα διαγράμματα των ε, στρωμάτων κάτω από την επιφάνεια, βάθος 800 3.000 μέτρα, Ε, τα πετρώματα από πάνω ε, περιέχουν στρώματα μη διαπερατά. Τώρα, είναι τεράστια η έκταση των κοιτασμάτων σχιστολιθικού. Βλέπετε εδώ την δυνητική περιοχή σε σχέση με την έκταση των συμβατικών κοιτασμάτων με κόκκινο και πράσινο που ίσως δεν το βλέπετε άμα κάθεστε πίσω. Αυτά τα συμβατικά κοιτάσματα είναι λίγα. Ε, αξιολογείται από την BGR και από, την, ε, και από το ερευνητικό κέντρο του Potsdam. Ε, δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για τη Γερμανία. Εν τω μεταξύ η EIA έχει ε, δώσει ότι η Γερμανία έχει 230 δις τετραγωνικά μέτρα ανακτήσιμα ε, σε σχιστολιθικό. Ε, οι μη συμβατικές πηγές είναι 40 φορές παραπάνω από την ετήσια παραγωγή σήμερα. Βλέπετε εδώ τους μεγάλους παίκτες που είναι η Πολωνία, η Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία Βλέπετε εδώ τα συμβατικά αποθέματα ε, είναι 4.500 ε, ε, δισεκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα. Είναι φυσικό αέριο σε πετρώδη σχηματισμούς με υψηλή αντίσταση στη ροή κάτω από τον ορίζοντα του πόσιμου νερού, 800 με 3.000 μέτρα. Ε, τα πετρώματα πάνω είναι μη διαπερατά και το δυναμικό είναι μεγαλύτερο από τα αποθέματα που είναι τώρα γνωστά. Επόμενο, πάμε στην ανάπτυξη. Ε, ε, έχουμε φρεάτια για να το αποκτήσουμε που συνδέουν την επιφάνεια με το κοίτασμα. Ε, έχουμε αγωγούς, χάλιβα και του συγκολούμε με ένα δακτύλιο. Ε, αυτός αυτό είναι ο σχεδιασμό ελέγχεται η ποιότητα με τεστ δοκιμασίες πιέσεως και ε, CBL ε, ο κύριος Χάουαρθ έδειξε κάποια τέτοια στοιχεία. Το αέριο μπορεί να πάει στον ορίζοντα ήμουν είδατος, αν η συγκόλληση είναι λάθος και αν και το κέλυφος είναι λάθος. Ε, ρογμάτωση χρησιμοποιείται για, για ε, σωστή ρογμάτωση, υδρολογική ρογμάτωση. Η τεχνολογία δεν είναι, και, ε, δεν είναι αγνωστή από το τέλος της δεκαετίας του 40. Ε, έχουμε ε, και σε αυτή την εικόνα εδώ συμβατικό φρεάτιο που έχει δύο πτερίγια σαν πεταλούδα και βλέπετε και τη διαφοροποίηση της ρογμάτωσης, της μεθόδου ρογμάτωσης για το ε, σχιστολιθικό αέριο που έχει αναπτυχθεί. Για, το για να μπορεί το σχιστολιθικό να γίνει ανακτήσιμο θα πρέπει να έχουμε μεγάλες ρογμές, σχισμές, ε, χρειάζεται να διοχετεύσουμε υψηλότερους, μεγαλύτερους όγκους νερού, 20.000 κυβικά, είναι πολλά όμως. Στη Γερμανία δεν έχω δει φρεάτια που χρησιμοποιούν τόσους μεγάλους όγκους νερού. Οι ρογμές δεν είναι καινούργια στη Γερμανία. Στη Γερμανία μετά από την αρχή της δεκαετίας του 60 περίπου 300 φρεάτια ε, αντιμετωπίζονται με ρογμάτωση ε, μεγάλες ρογματώσεις έχουν γίνει για να πάρουμε το μη συμβατικό συμπαγές αέριο. Ε, στις ΕΠΑ οι επιτυχίες ε, στηρίχθηκαν στη τεχνολογία υδρορογμάτωσης. 35.000 φρεάτια υπάρχουν στις ΕΠΑ το 2005 και η παραγωγή ήταν 17 δις κυβικά μέτρα το χρόνο. Η παραγωγή αρχικά περιορίζονταν στη ΣΥΠΑ σε ε, συγκεντρώσεις ε, διαφορετικές. Τώρα χρησιμοποιούνται σύγχρονες ε, τεχνολογίες ρογμάτωσης μαζί με την οριζόντια γεώτρηση, οριζόντια τεχνολογία, οριζόντια τεχνολογία και των πολλαπλών ρογματώσεων είναι καινούργιες. Βλέπετε εδώ πώς λειτουργεί σε κινούμενο σχέδιο. Εδώ βλέπετε ε, τα στοιχεία ε, από κοίτασμα στη ΣΥΠΑ. Το σχιστολιθικό ελασματοποιείται, ε, είναι εύθραυστο, εύθρυπτο, έχει πολλές ρογμές, σχισμές, έχει πόρους, ρηγματώνεται θα πρέπει να υπάρχει σύστημα ρογμάτωσης ε, ε, μεγαλύτερο από το φυσικό ή θα πρέπει να δημιουργείται. Αυτό το βλέπετε εδώ, βλέπετε εδώ τον σχιστολιθικό άργυλο και τα μικρότερα κομμάτια. Έχουμε εδώ το υγρό ρογμάτωσης που ακολουθεί τις ε, σχισμές και τις ρογμές στο σχιστολιθικό, στη σχιστολιθική άργυλο και μεταφερούμε το αέριο από το συστολιθικό με ε, διάχυση. Το αέριο μετά αφαιρεί, ε, διοχετεύεται. Η τεχνολογία, εξέλιξη της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται στη ΣΥΠΑ, τη βλέπετε εδώ σε αυτή την εικόνα. Εδώ βλέπετε 15 χιλιόμετρα Βλέπετε εδώ την ε, περιοχή που είναι πέντε φορές το μέγεθος έκτασης του Λουξεμβούργου, πενταπλάσια από το Βέλγιο. Ε, αυτό είναι το Barnett Shale, 10.000 ε, φρεάτια μέχρι το 2008. Εδώ βλέπετε πρώτα μέχρι το 2000, εδώ μέχρι το 2000, τα κατακόρυφες γεωτρήσεις μέχρι το 2000 ε, ήταν ε, λοξές, από το 2000 μετά ήταν οριζόντιες ε, και καμιά φορά γίνονταν πολλοί πλευρές Τώρα γίνονται multifrac, πολλαπλές ρογματώσεις σε πολλαπλά φρεάτια. Εδώ ε, μια περιοχή που περιέχει ε, φρεάτια της ίδιας κλίμακας που είδατε και πριν, αλλά η περιοχή εδώ είναι η Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, όπου περίπου 90.000 φρεάτια άνοιξαν συνολικά, με κίτρινο είναι πιο ρηχά, αλλά έχουμε μεγάλη πυκνότητα γεωτρήσεων και στη Γερμανία. Εδώ το κλειδί για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις είναι να μειώσουμε το κόστος, γιατί η μείωση του κόστους είναι το κλειδί. Ε, το κόστος για την κατασκευή ε, κυριαρχεί. Για τα, ε, πρέπει δηλαδή να μειωθεί το ε, κόστος κατασκευής των φρεατίων και της τεχνολογίας ρογμάτωσης. Αυτό για την ανάκτηση ενέργειας, όχι μόνο για το συστολιθικό αέριο. Χρειάζεται να μειωθεί το κόστος. Εδώ κάποιοι στόχοι... Εδώ ε, η δημιουργία σχισμών εξετάζεται και είναι μια καλά τεκμηριωμένη, καταξιωμένη τεχνολογία, εδώ και 60 χρόνια χρησιμοποιείται. Η περιβαλλοντική συμβατότητα πρέπει να υπάρχει παντού σε όλα τα μέτρα. Ε, το πέτρωμα από πάνω ε, θα πρέπει να περιέχει φραγές στη ροή το υγρό θα πρέπει από, από κάτω προς τα πάνω, πρέπει να έχει διαφορά πιέσεως για να γίνει αυτό, πρέπει να αυξάνεται η πίεση στο πέτρωμα, στο σχηματισμό, από όπου διαφεύγουν σε υψηλότερα στρώματα τα ύδατα, το υγρό. Θέλουμε να μειώσουμε την πίεση όμως εμείς, γιατί θα πρέπει να ανεβαίνει προς τα πάνω το υγρό στα ε, υπερκείμενα στρώματα. Θα πρέπει να είναι η σύνδεση καλή με την, ε, το κοίτασμα. Οι σχισμές, οι θα πρέπει να, να ε, περιέχονται μέσα σε συγκεκριμένο χώρο. Θα πρέπει το υγρό να είναι συμβατό με το περιβάλλον και ο όγκος του υγρού από τη ρογμάτωση πρέπει να μειώνεται. Μπορούμε να ξαναχρησιμοποιήσουμε το υγρό ρογμάτωσης από το ένα φρεάτιο στο άλλο. Η σύνθεση του υγρού φαίνεται εδώ, 90% είναι νερό, περίπου 9% ε, προπάνιο και 0,5% πρόσθετα, σύμφωνα με μια δημοσίευση της SPE. Υπάρχουν άνθρωποι που ε, ε, ισχυρίζονται ότι τα γνωρίζουν αυτά, πάντως ε, δεν είναι το δηλητηριώδες κόκτέιλ που περιγράφουν οι αντίπαλοι αυτή τη τεχνολογία στη Γερμανία. Χρησιμοποιούνται πρόσθετα που δεν είναι υψηλή τοξικότητας, ούτε είναι σπάνιες ουσίες, αλλά είναι γνωστές από συνήθεις άλλες χρήσεις. Ε, μέσα από την καθημερινή μας ζωή. Και τα βλέπετε εδώ τα παραδείγματα. Ε, όμως η βιομηχανία θα πρέπει να ψάξει να βρει και άλλες διαδικασίες που θα χρησιμοποιεί λιγότερες πρόσθετες ουσίες. Και στη Γερμανία μέχρι τώρα κατά το παρελθόν δεν χρησιμοποιούσαμε ε, αυτό το ε, ιδιωτικό νερό που χρησιμοποιείται, το slick water που χρησιμοποιήθηκε αλλού στη δεκαετία του 90 και του 80 και που μας επιτρέπει να μειώσουμε όμως τον αριθμό των πρόσθετων ουσιών όπως και τη συγκέντρωσή τους. Και αυτό φαίνεται εδώ. Αυτό στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί slick water. Αποτύπωμα θα πρέπει απάνω τα στρώματα να έχουν ε, κάποια φραγή ε, ε, στη ροή. Πρέπει να μειώσουμε το αποτύπωμα και αυτό μπορεί να γίνει και με τεχνολο... καινοτόμη... καινοτόμο ανάπτυξη της υποκείμενης επιφάνειας. Αυτό χρειάζεται και στην Ευρώπη. Θα πρέπει να πάμε από τα κατακόρυφα φρεάτια στα πολύπλευρα φρεάτια τα οποία ε, ρογματώνονται πολλές φορές και ελπίζομαι ότι στο τέλος θα έχουμε μια παρόμοια εικόνα ε, όπου από το ένα σημείο μπορούμε να ε, κάνουμε παροχέτευση πολλών χιλιόμετρων συστολιθικού αερίου. Ε, περιβαλλοντική συμβατότητα, ασφαλής ε, κατασκευή των ε, ρογματώσεων και των φρεατίων για να υπάρχει ανάσχεση των υγρών και αερίων από εκεί, ε, θα πρέπει να υπάρξει βελτίωση της συμβατότητας των ε, υγρών και καινοτόμως τεχνολογία για να μειωθεί το αποτύπωμα. Ε, τώρα τα κοιτάσματα στην Ευρώπη συμβατικών αερίων είναι λιγότερα από 5.000 δις, 10 στην 9 τετραγωνικά μέτρα. τα κοιτάσματα του σχιστολιθικού είναι πολύ μεγαλύτερες από 15.000 δις και είναι 50 φορές μεγαλύτερα τα κοιτάσματα συστολιθικού από τα παραγόμενα ε, ε, και τα αξιοποιούμενα κοιτάσματα αερίου, συμβατικού αερίου. Ευχαριστώ. Θα δώσουμε το λόγο και στον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Εμείς πάντως πρέπει να τελειώσουμε στις 5.30. Τώρα πότε θα προλάβετε να μιλήσετε όλοι δεν γνωρίζω. ίσως ε, πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των ειδικών. Αυτό οι ομάδες πρέπει να το εξετάσουν στις ακροάσεις. Θα πρέπει να έχουμε μικρότερο αριθμό εμπειρογνωμόνων για να μπορούμε να συζητούμε. Εγώ δεν μπορώ να λάβω απόφαση, οι συντονιστές εν τη σοφία τους θα τα αποφασίσουν όλα αυτά. Εγώ κάνω την πρόταση μόνο. Και τώρα η κύριοι Πενουά... Α, συγγνώμη από την Κομισιόν, ο κύριος ε, Ρόζενστοκ και ο κύριος Βινουά, είπαμε. Θα μας μιλήσουν εν συντομία και μετά οι παρεμβάσεις να είναι του ενός λεπτού για να προλάβουμε να ακούσουμε και τις απαντήσεις των εμπειρογνωμόνων. Λοιπόν, ποιος θα αρχίσει. Εσείς έχετε συνηθίσει να μιλάτε γρήγορα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Είναι πολύ απλό το ερώτημα προς την Κομισιόν. Ε, τι κάνουμε σε αυτή την κατάσταση. Και μαζί με τον συνάδελφο από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλον θα σας παρουσιάσουμε δύο απαντήσεις. Ουσιαστικά τη μία από την πλευρά της ενέργειας και την άλλη από την πλευρά του περιβάλλοντος. Καταρχάς θα ήθελα να σας μιλήσω για την ασφάλεια του εφοδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι είχαμε πληγεί από πολλές κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Το φυσικό αέριο τομέας που ε, δημιουργεί κάποιες ανησυχίες ό,τι αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού για διάφορους λόγους. Πρώτα απ' όλα την μείωση της ε, εγχώριας παραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως ε, βλέπετε σε αυτό το γράφημα είναι σταθερή τα τελευταία 20 χρόνια και επιταχύνεται ο ρυθμός και αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερες εισαγωγές. Βλέπετε λοιπόν την εξάρτηση από τις εισαγωγές φυσικού αέριου που από το 58% το 2005 θα φτάσει στο 83% το 2030. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Το σχιστολιθικό φυσικό αέριο είναι φυσικό αέριο, φυσικά. Ε, εξελίσσουμε, αναπτύσσουμε μια χώρια αγορά, μια τοπική αγορά στον τομέα αυτό και στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση στην αγορά για αυτό το αέριο εφόσον προκύψει και αυτό το οποίο κάνουμε είναι να ολοκληρώσουμε πρώτα απ' όλα την εσωτερική αγορά ενέργειας και την υποδομή. Θέλουμε να έχουμε ένα καλό ε, δίκτυο ευρωπαϊκό και θα κάνουμε και τις προτάσεις μας ε, για την ε, ενέργεια που θα καλύπτει βέβαια όχι μόνο το φυσικό αέριο αλλά και τον ηλεκτρισμό κτλ. Συγκεκριμένα τώρα, ποιες δραστηριότητες υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε καταρχάς ότι στην Ευρώπη σήμερα δεν υπάρχει κάποια διαθέσιμη εκτίμηση του οικονομικού ανακτήσιμου δυναμικού, διότι έχουν αρχίσει μόλις οι ερευνητικέ γεωτρήσεις και τα αποτελέσματα βέβαια θα τα έχουμε τα επόμενα χρόνια. Επομένως, εμείς πρέπει να παρακολουθούμε τι συμβαίνει και να δούμε ποιες πρακτικές εμπειρίες όπως στην Πολωνία μπορούν να μας φανούν χρήσιμες. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών ε, ανέλαβε να εκπονήσει μια μελέτη της βιβλιογραφίας για τον οικονομικό αντίκτυπο. Θα είναι έτοιμη στις αρχές του επόμενου έτους, το 2012. Και ο στόχος μας είναι να δούμε τι λένε οι διαθέσιμες πηγές και πόσο αξιόπιστα είναι τα στοιχεία και βάσει αξιόπιστα στοιχεία και χρησιμοποιώντας ενεργειακά μοντέλα θέλουμε να δούμε ποιος μπορεί να είναι ο μελλοντικό οικονομικός αντίκτυπος. Και φυσικά υπάρχει ανάγκη όλα αυτά να τα μελετήσουμε σε μεγαλύτερο βάθος, γιατί και σύγκριση με το τι συμβαίνει σα είπα πρέπει να κάνουμε, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η κατάσταση εδώ στην Ευρώπη είναι τελώς διαφορετική. Η αγορά, οι τιμές, και τα οικονομικά είναι τελώς διαφορετικά. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε και τα νομικά. Έχουμε λοιπόν μια νομική μελέτη αναθέσει για τα ρυθμιστικά πλαίσια σε διάφορα κράτη-μέλη και θέλουμε να δούμε πώς αυτό σχετίζεται με το νομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς στην Επιτροπή εξετάζουμε την κοινωτική νομοθεσία. Έτοιμη στα τέλη του Οκτωβρίου θα είναι αυτή η μελέτη και έτσι θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε και να εκτιμήσουμε ακόμη περισσότερο ε, την ε, αντοχή αυτής της, της κοινωτικής νομοθεσίας σε αυτή την τεχνική της εξόριξης αερόπωσης στο Λιθική Άργυλο. Επίσης, θέλουμε να βρούμε καλές εφημιστικές πρακτικές που θα μπορούσαν να διαδοθούν με τη βοήθεια της Κομισιόν και έχουμε και το φόρουμ του Βερολίνου για τα ορυκτά καύσιμα. Συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο στο Βερολίνο. Υπάρχουν ομάδες εργασίες και εκεί παρακολουθούμε εκ του αυτά τα θέματα. Ο συνάδελφός μου από τη ΓΑΜΑ Περιβάλλον θα σας πει τώρα περισσότερα για το τι κάνουν αυτοί από τη δική τους πλευρά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο γρήγορο όσο ήσουν εσύ. Δύσκολο βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, συντομία να σας συνοψίσω ποια είναι τα δυνητικά περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με την ε, παραγωγή σχιστολιθικού φυσικού αερίου και τις ε, δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Καμαδέλτα Περιβάλλον. Ακούσαμε τις διάφορες παρουσιάσεις. Κατά βάση μιλάμε για συνδυασμό δύο αρκετά πολύπλοκων τεχνολογικών διαδικασιών, οριζόντια γεώτρηση και υδραυλική γεώτρηση, υδραυλική συγγνώμη ρηγμάτωση υψηλού όγκου. Μια νέα σχετικά τεχνολογία για την Ευρώπη τουλάχιστον, ακούσαμε την αμερικανική εμπειρία. Από περιβαλλοντική σκοπιά τώρα, αυτό το οποίο ακούσαμε σήμερα νομίζω μας δείχνει ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα Έχουμε τα ε, χημικά που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες και το ενδεχόμενο ρήπανσης, μόλυνσης. Έπειτα έχουμε το θέμα της διαχείρισης αποβλήτων και λιμάτων, ε, ίσως κινητοποίηση, ε, έκκληση κάποιων ραδιενεργών συστατικών ουσιών. Το θέμα επίσης της ακαιρεότητας κατάστασης των σωληνώσεων για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται και τα υλικά και επίσης κάποια γενικά ζητήματα κεραιότητα, στο θέμα του υδροφορου κάποιες επικαλύψεις ε, με περιοχές Natura του 2000, που κάτι, είναι κάτι εντελώς ευρωπαϊκό. Περιορισμένη η εμπειρία μας μέχρι στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι δραστηριότητες που έχουν αναλυφθεί μέχρι στιγμή στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και όπως και προλαλή η εμπειρία από τη Βόρεια Αμερική είναι δύσκολο να μεταφερθεί ε, στην ε, Ευρώπη, είμαστε από κύριο Βον αυτά. Υπάρχουν και κάποια κενά σε ό,τι αφορά την ενημέρωση, τις πληροφορίες που μπορούμε να έχουμε για το περιβάλλον. Και βέβαια οι αβεβαιότητες δεν είναι καθόλου ε, καλές ε, για να έχουμε και την αποδοχή της κοινή γνώμη. Θα πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν την βάση, τη γνωσιακή που έχουμε, να δούμε ποιες είναι οι πιθανές εκπτώσεις, ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και βάσει αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με τη σχετική τεχνολογική ε, γνώση της τεχνολογίας. Τι κάνουμε λοιπόν, συλλέγουμε στοιχεία. Συλλέγουμε πληροφορίες για να έχουμε μια συνεκτική εικόνα των κινδύνων και των επιπτώσεων. Παρακολουθούμε τις ε, επιστημονικές εξελίξεις, τις εξελίξεις στα διάφορα έργα και εντός και εκτός Ευρώπης. Καταγράφουμε ε, και προσπαθούμε να προσετεριστούμε κάποιους ε, επιστήμονες και διάφορους ε, οργανισμούς για να έχουμε και περισσότερες πληροφορίες και από αυτούς. Αν δείτε συγκεκριμένα στη διαφάνεια, έχουμε τη λεγόμενη desk study, επιτραπέζια μελέτη, βιβλιογραφική μελέτη που θα μας δώσει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε τους πιθανούς κινδύνους για το περιβάλλον και για την ε, δημόσια υγεία, να δούμε τι γίνεται με τις μεθόδους της ρωμάτωσης και βάσει των πληροφοριών που θα έχουμε στη διάθεσή μας θα δούμε αν μπορούμε να προτείνουμε μέτρα διαχείρισης των κινδύνων. Και από τις μικρότερες μελέτες ε, περιμένουμε τα πορίσματα το πρώτο τρίμηνο του επόμενου χρόνου. Έπειτα, ένα δεύτερο και πιο μείζον ζήτημα είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ε, Χημικών Ουσιών, συγγνώμη, ΕΚΑ. Ο Ευρωπαϊκός λοιπόν, Οργανισμός Χημικών Ουσιών κλήθηκε να εξετάσει τους φακέλους ε, καταγραφής καταχώρησης στο REACH ε, των ουσιών αυτών που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν ε, στις επιχειρήσεις εξόριξης ε, συστολιθικού φυσικού αερίου και να δούμε και κάποιες βασικές λέξεις που θα εμφανίζονται. Με φάση λοιπόν αυτή την μελέτη των keywords που κάναμε, φαίνεται ότι στους φακέλους αυτούς δεν υπάρχουν αναφορές σε τέτοια keywords μία, ένα, τρία συμπεράσματα είναι πιθάνα. Το πρώτο, ότι οι ουσίες που ψάξαμε να βρούμε δεν είναι αυτές που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος ή αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από τους διάφορους φορείς. Άρα θα πρέπει να δούμε τελικά τι ουσίες χρησιμοποιούνται. Δεύτερο συμπέρασμα πιθανό, οι ουσίες που χρησιμοποιούνται είναι μένει σωστές, αλλά είναι κάτω του ορίου, ε, κάτω, του ορίου καταγραφής, καταχώρησης, άρα σε χαμηλές ποσότητες. Και τρίτη ε, πιθανότητα είναι ότι χρησιμοποιούνται αυτές οι ουσίες και πάνω από το κατόφλι, πάνω από το όριο, αλλά τα σενάρια έκθεσης δεν περιλαμβάνουν κάποια πληροφορία για αυτές τις ουσίες. Δηλαδή υπάρχει ανεπάρκεια στοιχείων, οπότε και φορείς ε, που αναλαμβάνουν την ε, γεώτρηση αυτή, την εξόρυξη του φυσικού αερίου όπως και δεν θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τους ενδεχόμενους κινδύνους, δεν θα έχουν τα τα στοιχεία, άρα πρέπει να έχουμε παραπάνω keywords που θα δώσουμε στην ε, έρευνα για αναζήτηση. Επίσης, στο Κοινό Κέντρο Ερευνών ζητήθηκε να μας, ζήτησαμε να μας υποστηρίξει με κάποιες ποσοτικές μελέτες βάσει ενός μοντέλου χωρικού χαρακτήρα, δηλαδή εξετάζονται ξεχωριστά κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί ακούσαμε ότι πολλά εξαρτώνται από τη γεωλογία, τις γεωλογικές συνθήκες, τα γεωλογικά χαρακτηριστικά του εδάφους. Δεν μπορούμε να προβούμε σε γενικόλογες διατυπώσεις. Θέλουμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι απαιτήσει ό,τι αφορά το νερό και τη γη. Και επίσης με την Αμερικανική ε, EPA και σε συνεργασία και με άλλες γενικές διευθύνσεις ανταλλάσσουμε πληροφορίες γιατί οι EPA στις είπα, κάνουν ε, πολλές αναλύσεις εκεί. Τέλος, νομική ανάλυση. Το περιβαλλοντικό κεκτημένο ισχύει σε όλα τα σχέδια εξορρόξης συντρογών ανθράκων, άρα τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίσουν την πλήρη συμμόρφωση προς όλες τις σχετικές οδηγίες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκτιμήσει επίσης το κατά πόσον πράγματι εφαρμόζεται το, κοινωτικό, το περιβαλλοντικό κοινωτικό κεκτημένο με βάση πληροφορίες που έχουμε. Άρα, λοιπόν, για να καταλήξουμε μπορούμε να πούμε ότι Καταρχήν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σαφέ συμφέρον ε, να βασιστεί σε χώρε ενεργειακέ πηγέ. Θα μπορούσε το συστολικό φυσικό αέριο να εξασφαλίσει την ε, ασφάλεια, μάλλον να συμβάλλει στην ασφάλεια του εφοδιασμού. Βέβαια θα αυξηθούν οι εισαγωγέ από ό,τι φαίνεται, αλλά σίγουρα θα βελτιωθεί η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου, αν θέλετε. Και αυτό είναι ενδιαφέρον για την Ευρώπη. Βέβαια, το φυσικό αυτό αέριο θα πρέπει να βρει τη θέση του στην αγορά, θα πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμο δηλαδή, και βέβαια να δούμε και τις δυνητικές ε, μελέτες επιπτώσεων και κινδύνων. Όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα λέμε πολύ σοβαρά υπόψη τους ε, οι αρχές αλλά και οι φορές εκμετάλλευσης. Είδαμε ότι πρέπει να βελτιωθεί η κατάσταση και σε ό,τι αφορά τις γνώσεις και, και σε ό,τι αφορά την ε, αξιολόγηση των κινδύνων. Επίσης και οι πολίτες θα πρέπει ε, να ε, δίνουν τη γνώμη τους. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν διαβούλευση, ενημέρωση των πολιτών ήδη από αρκετά πρώιμο στάδιο. Και εάν οι τεχνολογίες αναπτύσσονται και φαντάζομαι ότι σίγουρα θα αναπτυχθούν ακόμη περαιτέρω και αν ξεκινήσει εμπορική παραγωγή θα έχουμε διαφορετική κλίμακα σε μερικά χρόνια. Σήμερα λοιπόν πρέπει την διερευνητική αυτή φάση, τη δοκιμαστική φάση, να την αξιοποιήσουμε για να δούμε κατά πόσον χρειάζεται βελτίωση το ρυθμιστικό πλαίσιο. Αν πρέπει να ε, προετοιμαστούμε για τη μελλοντική εμπορική παραγωγή στο μέλλον δεν θα είναι την επόμενη τριετία από ό,τι φαίνεται. Μάλλον το 2020 είναι ένας πιο πιθανός χρονικός ορίζοντας. Το είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έτσι έχουμε και χρόνο να μελετήσουμε την κατάσταση και να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα, να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να υπάρχει ασφάλεια. Εμείς ως Επιτροπή θα παρακολουθούμε όλες τις εξελίξεις, όπως το ε, έχετε καταλάβει και εσείς φαντάζομαι, για να έχουμε το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο αλλά και σε κατάλληλα επίπεδα ασφάλειας, υψηλά επίπεδα ασφάλειας, κάτι που αναμένουν όλοι. Και επίσης και ο κλάδος, η βιομηχανία θα πρέπει να αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή για να βελτιώσει τις τεχνολογίες και τις ε, πρακτικές λειτουργίας. Πρέπει να παρακολουθούμε εκ του και στην κατάσταση, αυτό είναι πολύ απαραίτητο, αλλά δεν θα πρέπει να κάνουμε βεβαιασμένες κινήσεις, ε, γιατί αυτό δεν θα μας έδινε τη δυνατότητα να βρούμε σωστές λύσεις για κάποια ζητήματα που ενδιαφέρουν ε, πάρα πολύ την κοινή γνώμη, όπως είναι η ασφάλεια του εφοδιασμού και η εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Ένα λεπτό. Κύριο Σιμάνσκι πρώτος. Ευχαριστώ. Συμφωνώ. Είναι χρονοβόρος η διαδικασία αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είναι πολύ ενημερωτική. Χάρηκα που ήρθα ιδιαίτερα σε σύγκριση με την χθεσινή εκδήλωση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος που δεν ήταν τόσο ενημερωτική, ήταν πιο συναισθηματική, συναισθηματικά φορτισμένη. Τώρα, για το αποτύπωμα εκπομπών έχουμε πολλές πληροφορίες. Ακούμε το φυσικό αέριο και το συστολιστικό ε, κατά 50% δημιουργεί ε, λιγότερες εκπομπές. Ε, είναι σημαντικό αυτό ε, και για την Πολωνική και άλλες οικονομίες που εξαρτώνται από τον άνθρακα. Απ' την άλλη ο καθηγητής Χόουαρθ μας έδωσε την πληροφορία πολύ τρομακτική ότι το συστολιστικό έχει χειρότερο αποτύπωμα εις ό,τι αφορά ε, ε, χειρότερο από τον άνθρακα. Γιατί, γιατί υπάρχουν τέτοιες μεγάλες διαφορές στους υπολογισμού και στι αναλύσεις. Η καθηγητά Χόβαρθ, χρησιμοποιήσατε ένα χρονικό ορίζοντα διαφορετικό από τις IPCC ή χρησιμοποιήσατε το άνισμα ή ένα επίπεδο διαρροής που είναι συνηθισμένο στη Ρωσία αλλά όχι στην Ευρώπη τόσο πολύ. Γιατί στην Ευρώπη έχουμε τρεις φορές λιγότερες διαρροές ε, από τους αγωγούς από τη, στη Ρωσία. Δηλαδή γιατί, πού οφείλονται αυτές οι τεράστιες διαφορές στους υπολογισμούς σας. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα. Ε, Χωρίς μικρόφωνο. ακούσαμε διαφορετικά πράγματα. Εγώ είμαι ευγνώμων που θα τα λάβει όλα υπόψη η Κομισιόν όμως. Θα δει διαφορετικές πηγές και όλα αυτά θα τα ε, δει όπως ε, χτες ένα ε, ίδρυμα παρουσίασε στοιχεία στην Επιτροπή Περιβάλλοντων και είπα να γίνει μορατόριουμ γιατί όλα αυτά είναι πολύ επικίνδυνα για το περιβάλλον και την υγεία κλπ. Ενώ εσείς τώρα από ό,τι κατάλαβα είσαστε μέσα σε αυτή τη διαδικασία, μετράτε, κοιτάτε και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό. Επίσης έχουμε μεγάλη ε, διαφοροποίηση γεωλογική στα, στα πετρώματα, στα κοιτάσματα στην Ευρώπη. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα δεν μπορεί να γίνει μία και μόνο μέτρηση και να εφαρμοστεί μία και μόνο λύση όταν είναι τόσο διαφορετικά τα δεδομένα. Και αυτό είναι ερώτηση και προς τον Πρόεδρο. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δεν μπορούν να συνεργαστούν για να υπάρξει μια εκτίμηση για το σχιστολιθικό αέριο, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες ε, μετρήσεις και ε, μεθόδους. Στον πολωνικό τύπο αναφέρεται ε, επανειλημμένα μια φράση που θέλω να μου να την δούμε και να την επιβεβαιώσετε. Τελειώνουνε. Ο Γερμανός Επιτρόπος Σέτιγκερ είπε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου θα αντιπροσωπεύει πρότυπα Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξόριξη. Δεν διευκρίνησε αν θα είναι ε, κανονιστικά πρότυπα ή άλλα πρότυπα θα παρουσιάσει, όχι θα την προσωπεύσει, με συγχωρείτε, θα παρουσιάσει τα πρότυπα η Επιτροπή του χρόνου. Ευχαριστώ κύριο Ρότε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι καλό που αντιπαρατηθέμεθα με αυτό το θέμα. Ο κύριος Γκρότε ε, το παρουσιάσαμε άσπρο μαύρο, αλλά κάπου στο μέσον είναι η αλήθεια. Ε, ακούσαμε διαφορετικές απόψεις στη, στον Τάμε, την εκλογική μου περιφέρεια στην κάτω ε, Σαξονία. Ε, ε, πρωτοέγινε η ρογμάτωση το είπε ο κ. Ράινικεν, 40.000 ε, διαφορετικά χημικά πέρασαν ε, στο έδαφος και κανείς δεν γνωρίζει με ποια μορφή, ποια χημικά ε, πέρασαν στο έδαφος. Λίτρα, 24.000 λίτρα μόνο. Και οι δήμαρχοι αυτά δεν τα βλέπουν με καλό μάτι βέβαια. Η πρώτη προσέγγιση ήταν καλή, ο Πολωνός ε, ε, ομιλητής ε, που είπε ότι μιλάμε με τον κόσμο εκεί, με τις κοινότητες. Όταν θέλουμε να εισάγουμε μια νέα τεχνολογία πρέπει να γίνει σωστή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των διαφόρων πολιτικών επιπέδων και ανταλλαγή πληροφοριών. Ε, νομοθεσία πλαίσιο, η οδηγία πλαίσιο, πώς πρέπει να εφαρμοστεί, να προσαρμοστεί, τι πρέπει να περιμένουμε από την Κομισιόν σε ό,τι αφορά τα χημικά, τι γίνεται και αν είναι δυνατόν να μας το πούν οι ειδικοί, να μην χρησιμοποιούνται χημικά καθόλου, γιατί υπάρχει μεγάλη δυσφορία σχετικά με το θέμα αυτό και υπάρχουν και πρωτοβουλίες πολιτών κατά των χημικών αυτών. Ε, εδώ ε, σε αυτή την περιοχή το κόμμα του κυρίου Λάγκεν έχει την πλειοψηφία ε, και ίσως θα έπρεπε να ασχοληθούν με το θέμα αυτό γιατί τόσα πολλά χημικά να περνούν στο υπέδαφος. Υπάρχουν πολλοί δήμαρχοι ε, από το κόμμα του κυρίου Λάγκεν στη Γερμανία μου φαίνεται η πλειοψηφία. Τέλος πάντων. επόμενη ερώτηση ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ το συσυλλητικό αέριο θα μπορούσε να συμβάλλει στην ασφάλεια της, του εφοδιασμού, αν και οι εισαγωγές μάλλον θα αυξηθούν. Δηλαδή, δεν μπορούμε στην Ευρώπη να αξιοποιήσουμε πολύ και να εκμεταλλευτούμε το συσυλλητικό αέριο. Αν αποφασίσουμε για περιβαλλοντικούς ε, λόγους ή λόγους κόστους να μην προχωρήσουμε στο συστολιθικό στην Ευρώπη, αυτό πώς θα επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, την ασφάλεια του εφοδιασμού και αν απορρίψουμε επίσης την παραγωγή στην Ευρώπη του συστολιθικού αερίου, θα απορρίψουμε και τις εισαγωγές του συστολιθικού από τη ΣΥΠΑ για παράδειγμα που χρησιμοποιούν όμως παρόμοιες μεθόδους με τις δικές μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόνικ. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ έχω ερωτήσεις ε, για τον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν για τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Εσείς Αναφερθήκατε στο ότι θα υπάρξει νομοθεσία, νέα νομοθεσία. Μα έχετε, όπως είπε και η κυρία Μπομπίνσκα, κάτι στο νου σχετικά. Δέστε τι έγινε στο Μεξικό. Έχετε κάτι κατά νου επίσης και για την εκμετάλλευση των offshore εγκαταστάσεων στην Βόρεια Θάλασσα. Επίσης, τι έκανε η Κομισιόν για το Nord Stream, δεν κούνησε το δαχτυλάκι της. Είχε ζητήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνει μια περιβαλλοντική μελέτη στη Βαλτική θάλασσα για το Nord Stream, ξέροντας ότι υπήρχαν προβλήματα βλαβών στο βυθό της Βαλτικής. Και δεν μας απάντησε ποτέ η Κομισιόν, δεν έκανε ποτέ τίποτα. Gut. Danke sehr, Ευχαριστώ, e, Pan Ευχαριστώ πρόεδρε. Εσείς ήσασταν ιδιαίτερα αισιόδοξο για την διοχέτευση του σχιστολιθικού αερίου στην Αμερικανική αγορά. Χαίρομαι πάρα πολύ όμως με την τοποθέτηση του εκπροσώπου της Κομισιόν που λέει ότι θα πρέπει να εργαστούμε γύρω από το νομοθετικό πλαίσιο και να λάβουμε υπόψη μας τις επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες εργάζονται στην ευρωπαϊκή επικράτεια και αγορά. Τώρα ακούγοντας εδώ τον πρόεδρο πρέπει να σας πω ότι στην Πολωνία μας παρακολουθούν από κοντά. Και η περίοδος όπου βρισκόμασταν ακόμη σε γεωλογική απογραφή έχει εκπνεύσει τρία-πέντε χρόνια. για να μπορέσουμε πλέον να έχουμε τα απαραίτητα για την Ευρώπη στοιχεία και όχι για την Αμερική. Θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση. Θέλετε να παρέμβετε. Ε, ένα λεπτό όμως. Παρακαλώ. Από σήμερα το πρωί ήμασταν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όπου είχαμε τις, ε, μας παραδόθηκαν οι σχετικές εκθέσεις για τις υδραυλικές εξορίξεις. Λοιπόν, στη Γαλλία είχαμε ένα μορατόριο, πάγωμα, διότι ζήτησαν οι πολίτες να απαγορευτεί ή υδραυλική ρηγμάτωση, διότι αυτό είχε επιπτώσεις και στην ποιότητα του αέρος και στην ποιότητα του ύδατος. Τώρα αυτοί που θα εκμεταλλευτούν αυτές τις, ε, αυτά τα κοιτάσματα θα μπορέσουν να έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο είχαμε κενά για τις ε, κοινοτικές ρυθμίσεις και για τις μελέτες επιπτώσεων. Έχουμε 500 κυβικά τη μέρα παραγωγή φυσικού αερίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με σχίστολιθικό φυσικό αέριο. Επίσης, τι γίνεται με την υδρορογμάτωση και όλες τις ουσίες τις οποίες διοχετεύουμε. Τώρα, αν στην Πολωνία αποφασίσουν οι πολίτες ότι πρέπει να εκμεταλλευτούν τον, ε, το, το αέριο ποσχιστόλιθο δικαίωμά τους αλλά από τη μεριά της Ευρώπης είναι δικαίωμά της να εξα, υποχρέωσή της να εξασφαλίσει την ασφάλεια. Αν ήσασταν ε, όταν ήμουν ο Καραμπούλα θα τα είχατε καταλάβει όλα γιατί τα είπε για την Πολωνία. Καλά. Θα τα βρούμε αυτά μεταξύ μας. Ε, μην κάνουμε διαδικαστική συζήτηση. Δέκα λεπτά μας μένουν. Τέλος πάντων, θέλετε διαδικαστικά. Κύριε Λάγκεν, δεν μπορώ να σας τα απαγορεύσω. Μια παρατήρηση. Είναι κατάχρηση σε μία κροάση να έρχεται κάποιος από τηλεοπτικό συνεργείο, ε, τηλεοπτικό συνεργείο να μην κάνει καμία ερώτηση και να φεύγει μετά από λίγα λεπτά. Αυτά, μα γίνονται, πρέπει να ισχύουν για όλες τις ε, παρατάξεις και όλους τους συναδέλφους οι κανόνες έλευσης τηλεοπτικών ε, συνεργείων. Δεν μου είχαν πει ότι θα έρχονταν, δεν ξέρω καν ποιος ε, τους έφερε, δεν το ήξερα. Τέλος πάντων, άλλη φορά θα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ας κάνουμε νοικοκυρεμένη συζήτηση μέχρι να τελειώσει η ακρόαση. Και μετά θα συζητήσουμε μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα μεταξύ μας όπως πάντα. Ας δώσουμε το λόγο τώρα στους εκπροσώπους της Κομισιόν και τους ειδικού που ήρθαν για να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Ε, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, ποιος θα απαντήσει. Δεν είναι ανάγκη να λάβετε όλοι το λόγο. Κάποιοι ε, από τους προσκεκλημένους μας ε, που θέλουν να μιλήσουν μπορούν τώρα. Παρακαλώ. Μάλιστα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε κάποια ε, ερωτήματα που γνωρίζω για τις ε, δύο διαφορετικές, ε, τα δύο, τρία, δύο διαφορετικά νούμερα για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κλπ. Η μελέτη IEA αναφέρεται στη μελέτη από το Κορνέλ Υπάρχουν δύο βασικές διαφορές. Η μία είναι ο χρονικός ορίζοντας, 21% έτη για το μεθάνιο και τις εκπομπές μεθανίου. Όπως και άλλοι συγγραφείς πήραμε τα 100 χρόνια γιατί είναι η συνιστομένη περίοδος στην τελευταία μελέτη IPCC, IPCC του 2007 Σωστά είπε ο καθηγητής Χόαρθ ότι μπορεί να μην είναι ε, η καλύτερη επιστημονικά τεκμηριωμένη περίοδος και υπάρχουν ε, επιχειρήματα υπέρ του μικρότερου χρονικού ορίζοντα γιατί παραμένει το μεθάνιο τότε στην ατμόσφαιρα. Από την άλλη να πω ότι όλες οι χώρες που αντιπροσωπεύονται εδώ ε, αναφέρουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου στα Ηνωμένα Έθνη και όλες αυτές οι αναφορές στηρίζονται στη μελέτη IPCC και τα ισοδύναμα από εκεί. Αν θέλετε να αλλάξετε και μπορεί να αποφασίσει η IPCC να αλλάξει, ε, θα πρέπει η αλλαγή να γίνει για όλες τις πηγές εκπομπών μεθανίου, όχι μόνο για τις εκπομπές μεθανίου από το συστολιθικό αέριο που είναι μόνο ένα μέρος, ε, μια πηγή μόνο εκπομπών μεθανίου, υπάρχουν πολλές ε, λόγω της γεωργίας και άλλες πηγές εκπομπών μεθανίου. Αυτή είναι η πρώτη πηγή που διαφορά στον νούμερων. Η δεύτερη διαφορά οφείλεται στο ότι η ποσότητα μεθενίου που εκλείεται στην ατμόσφαιρα ανά μονάδα παραγωμένου μεθανίου και είπε καθηγη... Ε, αναφέρθηκαν ε, τα νούμερα, το PPA παρουσίασε ένα, μια τιμή ε, που είναι στο ενδιάμεσο. Εμείς μιλήσαμε την EPA, φαίνεται ότι αυτά τα 0,25 που αναφέρονται, είναι το χειρότερο σενάριο όταν όλο το μεθάνιο μέσα από την ε, διαδικασία παραγωγής ε, με υδραυλική ρηγμάτωση περνάει στην ατμόσφαιρα, οπότε αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, η χειρότερη τιμή. Ε, κάναμε εκτιμήσεις με την EPA για να καταλήξουμε σε μέσο αριθμό εκπομπών για τις ΕΠΑ και πάλι παίρνοντας στοιχεία από την EPA, αν χρησιμοποιήσουμε βέλτιστες πρακτικές και δεν γίνει ε, καύση σε λιχνία και δεν γίνει και ε, εξαέρωση, μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εκεί οφείλονται οι διαφορές. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να σχολιάσω λίγο είναι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην υδραυλική ρογμάτωση. Ε, υπάρχουν διάφορα ε, χημικά δύο κατηγοριών είναι πολυμερή. Είναι το slick water, η ρογμάτωση χρησιμοποιώντας αυτό τον τύπο, ε, πολυακρυλαμίτης, ε, γκορ, πολυμερή γκορ, κυταρίνης. Ε, μοιάζουν με τα πολυμερή όμως που χρησιμοποιούνται και στα τρόφιμα αν και η βιομηχανία δεν χρησιμοποιεί πολυμερή από, που χρησιμοποιούνται στα τρόφιμα ακριβώς, αλλά παρόμοια. Θα μπορούσαν να τύχουν επεξεργασία για να φτάσουν στο επίπεδο των πολυμερών που χρησιμοποιούνται στα πολυμερή. Επίσης θα πρέπει να προληφθεί η οξύδωση αυτών των πολυμερών. Ε, αυτό γίνεται σε πολλές άλλες, άλλους κλάδους της βιομηχανίας. Ο κύριος Χάουαρθ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σχολιάσω λίγο περισσότερο τις διαφορές μεταξύ των, της δικής μας μελέτης και άλλων. Το χρονοδιάγραμμα της ανάλυσης είναι μία διαφορά και σε ό,τι αφορά τα στοιχεία για τη διαρροή μεθανίου. Εκεί χρησιμοποίησαμε νομίζω τι καλύτερε διαθέσιμε πληροφορίε. Εξακολουθώ να το πιστεύω αυτό. Αν δείτε ότι είναι καλύτερε δηλαδή, αν δείτε τα στοιχεία εξαέρωση στην περίοδο του flowback, οι εκτιμήσει είναι χαμηλότερε από αυτή του Οργανισμού Προστασία του Περιβάλλοντο. Μία από τι βασικέ ε, βεβαιότητε που έχουμε είναι την παραγωγή ε, στη διάρκεια του χρόνου ζωή ενό φρεατίου, μια γεώτρηση. Ε, παραγωγής ενέργειας. Είναι πολύ λεπτός ο υπολογισμός και πολύ σημαντικός. Εμείς πήραμε επταετή κατά παραγωγή βάσει των δεδομένων από τα Βεάτια Μπαρνέλ και Μαρσέλ που νομίζουμε ότι είναι καλά τα στοιχεία ε, ενώ ε, η EPA χρησιμοποίησε κάτι ε, άλλο ως υπολογισμό. Φυσικά και υπάρχει αβεβαιότητα, είναι καινούργια η τεχνολογία και δεν μπορούμε να ξέρουμε λεπτομέρειες για την τεχνολογία αυτή, αλλά είναι πλήρης η αβεβαιότητα, δεν την έχουμε μόνο ε, είναι παντού. Τώρα, το IPCC και οι αρχικέ προσπάθειες ε, με την εκατονταετία ως χρονοδιάγραμμα στην συνθετική έκδοση 2007 εξακολουθούσε να λέει ότι χρειαζόμαστε μια βάση σύγκρισης ε, Είχαν λοιπόν επιλέξει την εκατονταετία, όμως ε, είπαν ότι θα πρέπει να προσέξουμε και την 20ετία ανάλυση και είπε η Κυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος ότι θα το ε, εξετάσει το δεχόμενο να περάσει στην 20ετία και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Εθνών το καλοκαίρι εξέδωσε μια έκθεση που λέει ότι οι κυβερνήσει θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο ε, την έκκληση θερμοκηπιακών αερίων όπως, όπως μεθανίου θέλουμε να μην υπάρξει ε, μεγαλύτερη υπερθέρμανση του πλανήτη αφενός και αφετέρου πρέπει να δούμε ε, και τα σενάρια που έχουμε για τις επόμενες δεκαετίες ό,τι αφορά την θέρμανση του πλανήτη. Πώς θα προστατεύσουμε δηλαδή ε, τον πλανήτη. Είναι σημαντικά και τα δύο χρονοδιαγράμματα και τα δύο τα εξετάσαμε, αλλά βλέποντας όλες τις μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, νομίζουμε ότι η μελέτη μας συνάδει με άλλες, λέγοντας ότι αν δούμε χρονοδιαγράμματα κάτω από 50 χρόνια, έχει πολύ κακό αποτύπωμα όσον αφορά την εκπομπή θερμοκηπιακών αερίων, το σχιστολιθικό φυσικό αέριο. Ευχαριστώ. Υπάρχει, φαίνεται, διαφορά στην αξιολόγηση των ε, στοιχείων αλλά και των δικτών που χρησιμοποιούνται για τις μετρήσεις. Θα είμαι σύντομος. Δύο ερωτήσεις πάνω στο ίδιο θέμα αφενός αν εφαρμόζουμε επιλεκτική προσέγγιση με την έννοια ότι μπορεί να είμαστε πιο αρνητικοί προς το σχιστολιθικό αέριο και από την άλλη αν υπάρχουν νομοθετικά κενά που πρέπει να πληρωθούν. Δηλαδή ε, έμεσα μπορεί ε, εκεί να μην δουλεύουμε αρκετά. Δεν κάνουμε επιλεκτική προσέγγιση, το περιβαλλοντικό κεκτημένο ισχύει για όλα τα έργα με υδρογονάνθρακε συμπεριλαμβάνοντα το σχιστολιθικό, αλλά όχι αποκλειστικά σχιστολιθικό. Τα κράτη-μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσει θα πληρούν απόλυτα την περιβαλλοντική νομοθεσία και υπάρχει ε, υπάρχουν παραδείγματα, είναι η οδηγία ΕΠΕ, για το, η οδηγία πλαίσιο για, το υδά, ε, για τα ύδατα, τη ΡΙΤΣ, η οδηγία για τα υπόγεια ύδατα. Αυτή τη στιγμή ε, είμαστε ε, στο στάδιο συλλογής πληροφοριών, παρακολουθούμε αυτά που συμβαίνουν, ε, πώς εξελίσσονται τα έργα, τα επιστημονικά έργα και πάνω στη βάση των πληροφοριών που συλλέγουμε θα αξιολογήσουμε αν υπάρχει ανάγκη να κάνουμε κάτι ακόμα ή αν είναι αποτελεσματικό το υπάρχουν και εκτιμένο. Και για να ε, ολοκληρώσω κι εγώ, κυρία ε, ε, Ολάρσκα, ίσως υπήρξε κάποια παρεξήγηση. Αναφέρθηκε στον επόμενο έτος. Αυτό θα το δει η Κομισιόν. Υπάρχουν πολλές κοινέ πληροφορίες στην Κομισιόν. Οι τρεις επίτροποι ε, συνεννοούνται και ο Επιτροπός Έτιγκερ παρακολουθούμε, αξιολογούμε την κατάσταση και πρέπει να υποβάλουμε προτάσεις αν υπάρχουν ενδείξεις ότι κάτι πρέπει να γίνει. Και βεβαίως δεσμευόμεθα και εμείς από εκτιμήσεις ε, επιπτώσεων ΕΠΕ και πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Όλα τα στοιχεία που ακούσαμε σήμερα το απόγευμα δείχνουν ότι χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση και αξιολόγηση, εκτίμηση της κατάστασης. Στον κύριο Κέλλη θέλω να πω ναι, οι καλύτερες υποθέσεις που έχουμε για το σχιστολιθικό αέριο είναι 5 με 10% της εγχώριας κατανάλωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή 500 BCM τώρα, οπότε κάνετε τον υπολογισμό σας, αλλά με την εξάντληση των ε, υπαρχών των κοιτασμάτων αερίου, ακόμα χρειάζεται να έχουμε περισσότερες εισαγωγές από ό,τι έχουμε τώρα. Ε, όπως είπα λοιπόν, η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου είναι απόλυτα ζωτική σημασία για την ασφάλεια εφοδιασμού και τον ανταγωνισμό αέριο προς αέριο που είναι κάτι που θέλουμε να διασφαλίσουμε. Ευχαριστώ, κύριος Ράινικε. Θα ήθελα να απαντήσω σε δύο ερωτήματα, αν κατάλαβα καλά. Ένα ερώτημα ήταν αν μπορούμε να συνεργαστούμε για την ανάπτυξη κοινών προτύπων και κανόνων. Φυσικά και συμφωνώ. Κανένα πρότυπο δεν είναι τέλειο, όλα επιδέχονται βελτίωσης. Και η ρογμάτωση για το φυσικό αέριο από σίγουρα είναι διαφορετική διαδικασία από αυτή που χρησιμοποιούμε για το συμβατικό αέριο. Και φυσικά θα πρέπει να βελτιώσουμε τα πρότυπα. Δεύτερο ερώτημα. Για τον Ντάμα στο Μίνουσελαντ. Δύο ερωτήσεις ουσιαστικά ήταν. Η πρώτη αφορούσε το κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα υδρορυγμάτωσης χωρίς χημικά. Στα γεωθερμικά φρεάτια η υδρορυγμάτωση ε, ε, γίνεται χωρίς χημικά. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσον αυτό μπορεί να λειτουργήσει και στην περίπτωση του σχιστόλιθου, θα πρέπει να το ελέγξουμε, να θα πρέπει να κάνουμε πειράματα. Και το δεύτερο υποερώτημα ήταν αν υπάρχουν άλλες τεχνικές διέγερσεις που δεν απαιτούν καθόλου υγρά, καθόλου ρευστά. Αν είχα, ξέρετε τώρα την απάντηση, αντί να είμαι στο πανεπιστήμιο και να εργάζομαι ως ερευνητής, θα είχα καταθέσει δίπλα με βρεσιτεχνία. αλλά δεν την έχω την απάντηση. Νομίζω ότι πρέπει να περάσουμε στην υδρορογμάτωση, στα water fracks, αλλά να μειώσουμε τον αριθμό των πρόσθετων ε, ουσιών και Επίσης να μειώσουμε και τις συγκεντρώσεις ακόμη περισσότερο. Και να δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Άλλο ερώτημα. Ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος διάλογος μεταξύ των εταιριών που κάνουν τις ε, δραστηριότητες αυτές και της ε, κοινότητας εν γέν. Κοιτάξτε, εγώ δεν συμμετέχω σε αυτά, αλλά από ό,τι μου λέει η κοινότητα, η ExxonMobil, παραδείγματος χάρη, έχει έναν διάλογο ε, θεσπίσει. Τώρα δεν ξέρω αν έχουν ε, ε έναν οικολόγο εκπρόσωπο ο οποίο ε, έχει επαφή με το τοπικό περιβάλλον, με την τοπική κοινωνία. Αυτό δεν το ξέρω ακριβώς. Αλλά αν υπάρχουν ζητήματα, αν παραμένουν προβλήματα, θα πρέπει να το δοκιμάσουμε, θα πρέπει να το ελέγξουμε. Αλλά από ό,τι έχω δει εγώ και είχα λάβει μέρος στο Βερολίνο σε μια παρόμοια ακρόαση που έγινε παρουσία κάποιων υπαλλήλων ε, ευρωβουλευτών, τι να σας πω, πρέπει να το δοκιμάσουμε. Δεν έχω δει κάτι καλύτερο από τη μάθη που χρησιμοποιούμε μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο εκπρόσωπος της Πολωνικής Προεδρίας, δεν ε, είχα αντιληφθεί ότι θέλατε κι εσείς να ε, μιλήσετε. Παρακαλώ, η Πολωνική Προεδρία έχει το λόγο. Hi, uh, my name Mike Griffin. I'm from Μάικ Γκρίφιν από το Πανεπιστήμιο αναφέρθηκα ε, αναφέρθηκα ως ε, συμμετασχόν σε μία από τις ε, εκθέσεις που παρουσιάστηκαν. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. Εσείς είστε επιστή, ο επιστήμον. Ε, κάποιος μου είπε ότι ήθελε να μιλήσει ένας εκπρόσωπος της Πολωνικής Προεδρίας. Ποιος, είναι, ποιος εκπροσωπεί? Εμείς εκπροσωπούμε την Πολωνική Προεδρία. Έχουμε τον καθηγητή Γκρίφιν ε, που είναι εξέχων επιστήμων και αναφέρθηκε από τον καθηγητή Χάουαρθ. Γι' αυτό πιστεύομαι ότι στο πνεύμα αυτό της ε, ε, αξιόπιστη ε, ε, επιστημονική συζήτηση μπορούμε να παρουσιάσουμε κάποια στοιχεία αν δεν έχετε πρόβλημα για να πάρετε τις πληροφορίες που διαθέτουμε. Α, συγγνώμη, έχουμε καλέσει πραγματογνώμονες, οι ομάδες αποφασίζουν ποιος θα προσκληθεί και όποιος προσκληθεί έχει και δικαίωμα λόγου. Εδώ έχουμε έναν ακόμη επιστήμονα, ε, ο οποίος θα μπορούσε ίσως να διευκρινίσει κάποιο, αν, το παράθεμα αν αναφέρθηκε με λάθος τρόπο και να θέσει τα πράγματα σωστά. Αλλά δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο τώρα σε ε, ε, εμπειρογνώμονα. Αν θέλετε μπορείτε να συντάξετε μια επιστολή την οποία θα αναλάβω εγώ να διανύμω στους ε, συναδέλφους. Αν θέλετε να ε, θέσετε, ε, να διορθώσετε κάτι. Αλλά εδώ μπορεί να παρευρίσκονται και δέκα εκπρόσωποι επιχειρήσεων. δεν μπορώ σε κάθε παρόμοια περίπτωση να δίνω σε όλους το λόγο. Σας υπόσχομαι, εάν μου κάνετε μία διόρθωση και μου πείτε ότι κάτι δεν παρετέθη σωστά, ε, τότε εγώ θα αναλάβω τα σωστά στοιχεία να τα δώσω σε όλους τους συναδέλφους. Αυτό ως συμβιβαστική λύση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ όλους τους συμμετασχόντες. Ε, ε, ήταν κουραστική ακρόαση, η οποία όμως μας έδωσε πολλές πληροφορίες και δείχνει ότι σε πολλά σημεία θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίρνουμε πληροφορίες. Δεν, φτάσαμε, δεν είναι αυτό το τέλος μιας διαδικασίας. Λοιπόν, σε δύο-τρία λεπτά θα αρχίσει η συνάντηση των συντονιστών.